Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Από το ΕΛΚΑ και του ΣΑΛΔΕ έχω προτάσεις για διορισμούς στις αντιπροσωπείες. Θα δημοσιευτούν στα πρακτικά και αν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρχει ένσταση, τότε οι διορισμοί θα ισχύσουν ως επιβεβαιωμένοι. Επόμενο σημείο, κοινή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Εύρεση Τεχνίας έχουμε την έκθεση του κυρίου Ραπ Κάι για τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών του κυρίου Μπαλτασαρέ για τις, ε, ε, το ενιαίο καθεστώς προστασίας και του κυρίου Λένε δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές. Ο κύριος Κάι έχει το λόγο πρώτος για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε διακεκριμένοι και πολύ άριθμοι συνάδελφοι, πριν από λίγες εβδομάδες στην εκλογική μου περιφέρεια επισκέφθηκα σε μια, μια επιχείρηση υψηλής καινοτομίας και παρουσίασαν τις ευρασιτεχνίες τους. Και Αντέδρασα αυθόρμητα και τους ρώτησα τι γνώμη έχουν για το ενιαίο δίπλωμα στην Ευρώπη με ενιαία προστασία γιατί περί αυτού πρόκειται. Και μου απάντησαν αυθόρμητα δεν το χρειαζόμαστε άμεσα, δεν το χρειαζόμαστε σήμερα ή αύριο, το χρειαζόμαστε χτες, όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί την ε, ε, ε, ευρεσιτεχνία την έχουμε αλλά την προστασία δεν έχουμε και αυτήν δεν τη χρειαζόμαστε ε, αύριο, ή σήμερα, τη χρειαζόμαστε χθες. Το πρόβλημα όμως είναι αγαπητοί μου συνάδελφοι ότι μετά από μακρές συζητήσεις για το ενιαίο δίπλωμα και ο συνάδελφος Λένε θα μας τα πει περισσότερο καλά για την ιστορία του όλου θέματος διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρολίγο να ε, παρεμποδίσουν για ακόμη μία φορά τις εξελίξεις. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γιατί ήδη είχαμε επιτύχει κάποια αποτελέσματα μετά από σύντομες αλλά πολύ επικοδομητικές ε, διαπραγματεύσεις είχαμε με την Πολωνική Προεδρία ετοιμάσει ένα πακέτο στο οποίο είχαν συμφωνήσει όλοι. Και μάλιστα η Πολωνική Προεδρία μας έδωσε γραπτά τα αποτελέσματα και μας είπε ότι θα ψηφίσει το Συμβούλιο όπως είχαμε συμφωνήσει. Ένα σημείο έλειπε μόνο. Η έδρα, έδρα του κεντρικού τμήματος του δικαστηρίου. Και εκεί δεν είχαν συμφωνήσει. Αυτό είναι καθήκον του Συμβουλίου. Δεν συμφώνησαν λοιπόν, συμφώνησαν μετά, έκαναν αίτηση τρεις χώρες για να πάρουν την έδρα και ποια ήταν η συμβιβαστική λύση. Τρεις χώρες θα έπαιρναν την έδρα. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν έκαναν αίτηση 8, αλλιώς θα έπαιρναν και οι 8. Το πρόβλημα είναι όμως ότι συνδέθηκε αυτό με το προαπαιτούμενο ότι τα βασικά στοιχεία για τον κανονισμό θα έπρεπε να αποσυρθούν χωρίς να αντικατασταθούν από κάτι άλλο. Παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή λαμβάνει μια απόφαση που παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο Δηλαδή θέλει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγει από τη διαδικασία. Το Δικαστήριο θα πρέπει δηλαδή με, με, με τη βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να βγει απ' έξω. Δηλαδή, εδώ παραβιάζονται δικαιώματα. Αυτές είναι οι τρεις κόκκινες γραμμές. Και είπαμε ότι αν πρόκειται να συνεργαστούμε εμείς και να σας ακολουθήσουμε, γιατί βέβαια θα, το ε, Συμβούλιο ε, είχε πει ότι το ε, άρθρα 6 θα έπρεπε να αποσυρθούν. Και σε μας δεν είπε τίποτα, αλλά για το Συμβούλιο Υπουργών ε, θα έπρεπε να το προσέξει. Εκεί λοιπόν υπήρχε πρόβλημα. Για να διατηρηθούν λοιπόν τα προσχήματα και για να συνεργαστούμε εμείς είπα ότι δεν μπορούμε να διαγράφουμε τα άρθρα 6 με 8 χωρίς αντικατάσταση. Χρειάζεται μια σωστή αντικατάσταση. Και εδώ άσκησα πολύ σκληρή κριτική στο Συμβούλιο, εξαιρώντας όμως ρητά την Κυπριακή Προεδρία, η οποία πήρε την καυτή πατάτα την οποία έπρεπε να διαχειριστεί. Και το έκαναν με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Εμείς ως Κοινοβούλιο είπαμε όμως ότι έτσι πρέπει να είναι η συμβιβαστική λύση, αλλιώς δεν γίνεται τίποτε. Και πράγματι αυτό ήταν το αποτέλεσμα, πετύχαμε αυτό που θέλαμε και πρέπει να πω ότι δεν είναι η ωραιότερη λύση που επιτύχαμε, αλλά είναι μια ε, συμβατή ε, λύση που έλαβε υπόψη τις τρεις κόκκινες γραμμές. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε, να ψηφίσουμε και να το αποφασίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο επόμενος ομιλητής για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Μπαλτασαρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, με τη σημερινή ψηφοφορία ολοκληρώνουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο εδώ και 40 χρόνια έχει ξεκινήσει. Επιτέλους θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια αποτελεσματική μέθοδο προστασίας του συστήματος. Το σύστημα ως έχει σήμερα είναι ε, περίπλοκο, αβέβαιο νομικά, ανασφαλές νομικά και είναι κάτι που ε, επιβραδύνει τις διαδικασίες καινοτομία. Το να περάσει κανείς ένα δίπλωμα σε ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται άνω των 30.000 ευρώ, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείες το αντίστοιχο κοστίζει 1.800 ευρώ και ισχύει σε όλες τις πολιτείες το να διατηρήσουμε ένα δίπλωμα ευαισθητεχνία στην Ευρώπη εν τω μεταξύ κοστίζει έξι φορές περισσότερο από ό,τι στην Ιαπωνία ή τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και επειδή δεν υπάρχει μία ενιαία διαδικασία για όλες τις νομικές υποθέσεις, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πολλαπλά συστήματα νομικά, πολλαπλές νομικές δικαιοδοσίες και δεν υπάρχει μία ενιαία μορφή αντιμετώπισης. Αυτό δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση στην, στην ε, ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, παρεμποδίζει την καινοτομία η οποία παραμένει στατική και πολύ διασπασμένη. Λόγω λοιπόν αυτών των αρνητικών καταστάσεων έρχεται το νέο σύστημα το οποίο θα μειώσει το κόστος ε, και ε, το κόστος των μεταφράσεων θα είναι από 4 με 6.000 ευρώ θα, ε, δώσει, θα προσφέρει επίσης και την νομική βεβαιότητα η οποία απαιτείται. Εγώ ως εισηγητής προσπάθησα να διευκολύνω την είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της νομικής αυτής ρύθμισης. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ένα αντισταθμιστικό σύστημα του συνολικού κόστους των μεταφράσεων θα είναι διαθέσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καταθέτουν μια αίτηση ευρεσιτεχνία σε διαφορετική γλώσσα από αυτήν στην οποία, της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους. Σύμφωνα με την ίδια λογική, ο κανονισμός για, την, για το ενιαίο δίπλωμα τεχνίας ρυθμίζει επίσης και τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σχετικά τώρα ε, την μόνιμη αυτή συζήτηση που γίνεται για τα θέματα τα γλωσσικά. Να πω ότι το μεταβατικό, ε, ο μεταβατικός αυτός χρόνος των 12 ε, ετών οδηγεί θα έλεγα προς την αγγλική γλώσσα μέσω βέβαια της δυνατότητας μελλοντικών ρυθμίσεων. Να πω τώρα για τις συμβιβαστικές λύσεις που προτείνονται. Το θέμα δεν είναι εμείς να τονίσουμε την απαράδεκτη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο στάθηκε αρνητικά σε ένα θέμα το οποίο αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είχαμε δύο δρόμους, ή εμείς να προχωρήσουμε στη μάχη ανάμεσα στους διαφορετικούς θεσμούς ξεκινώντας μια δεύτερη ανάγνωση ή να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση η οποία θα επέτρεπε όμως την πραγματική δημιουργία μιας μορφής προστασίας του διπλώματος σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της ευαισθητεχνίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν. Ταυτόχρονα δίδονται εγγυήσει έτσι ώστε η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών να είναι εφικτή σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Νομίζω ότι σήμερα θα εγκριθεί το πακέτο για το ενιαίο δίπλωμα και θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα νομικά βέβαιο, ασφαλές, χαμηλού κόστους που να διευκολύνει τις μικρομεσαίες, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο επόμενος ομιλητής για τέσσερα λεπτά, ο κύριος Λένε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το δίπλωμα έβρεση τεχνίας είναι συζήτηση από τη δεκαετία του 70. Από τότε υπήρχε το αίτημα στην Ευρώπη να υπάρχει ενιαίο σύστημα για τις ευρεσιτεχνίες. Το 2001 τότε επίτροπος Μπόλκεστάιν έκανε συγκεκριμένη πρόταση για κανονισμό για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η πρόταση τότε απέτυχε λόγω των αντιπαραθέσεων στο Συμβούλιο διότι για τους χρήστες και όλους όσοι ε, ασχολούνταν με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν ε, είχε σημασία αυτό. Ε, υπήρχε πρόβλημα με, το, με τις γλώσσες ως επιτοπλίστων στα αγγλικά υποβάλλονται οι αιτήσει και οι έρευνες παρουσιάζονται στα αγγλικά. Δύο ακόμα γλώσσες παίζουν κάποιο ρόλο, οι υπόλοιπε στις ευρεσιτεχνίες δεν παίζουν σχεδόν κανένα ρόλο. Τότε έγινε η πρώτη απόπειρα λοιπόν και απέτυχε για αυτούς τους λόγους. Θυμίζω ότι ως εκπρόσωπος της Επινομικής Επιτροπής και κατά το παρελθόν συχνά Είχα κάνει ταξίδια σε πολλές χώρες ε, στον κόσμο και στην Κίνα και ξέρετε την αντιπαράθεση της Ευρώπης με την Κίνα για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Και πάντοτε ακούγαμε από τους Κινέζους πόσο οπισθοδρομικοί είμαστε εμείς στο θέμα αυτό. Και στην ενιαία αγορά δεν είχαμε νέο σύστημα ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό δείχνει πόσο κατεπήγον είναι επιτέλους να επιληθεί το πρόβλημα. Ε, έχουμε επίσης ένα σύστημα, το είπε ο κύριος Ράπκαη, που είναι καλό για τις μεγάλες πολυεθνικές, αλλά δεν εξυπηρετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα με ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, το οποίο θα μπορεί να επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο και έτσι πολλά μειονεκτήματα για τις μικρομεσαίες θα αποφεύγονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε μεγάλο ρόλο για το, πακέτο, για το πακέτο αυτό. Εμείς θυμίζω είμαστε που στην προηγούμενη θητεία πιέσαμε την Κομισιόν να χαράξει νέα στρατηγική και είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο Μπαρνιέ ο οποίος ε, τις δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας τις αξιοποίησε και τώρα υπέβαλε νέα πρόταση ή νέο πακέτο ως πρόταση ούτως ώστε επιτέλους μετά από μακρές συζητήσεις να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η συνθήκη της Λισαβόνας όντως μας έδωσε νέα βάση για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και μας δίνει και τη δυνατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας μέσω της οποίας επιτέλους καταφέραμε να ξεπεράσουμε το γλωσσικό πρόβλημα και να καταλήξουμε σε μια λύση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για, τα, το, θέμα, για το θέμα των διπλωμάτων. Το δικαστικό σύστημα που έχω να παρουσιάσω και είναι και το αντικείμενο της έκθεσής μου είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός της ε, νομικής δομής, ε, δικαιικής νομής. Θυμάστε ότι είχε αναλάβει το δικαστήριο να ε, εξετάσει το θέμα ενός κεντρικού συστήματος και δεν γνωμοδότησε υπέρ αυτού. Έδειξε σαφώς το δρόμο προς μια δικαιοδοσία η οποία είναι μεν υπερεθνική όπως στις χώρες Μπενελούξη για τη δημιουργία ενός συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αλλά ε, λειτουργεί ως εθνικό δικαστήριο σε σχέση με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα δεν έχουμε να αποφασίσουμε πάνω σε αυτό, γνωμοδοτούμε μόνο. Ε, όμως ε, θα πρέπει να δεχτούμε ότι όλοι ελήφθησαν υπόψη και καταφέραμε εκεί το εξής. Εκεί όπου υπάρχουν αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη για θέματα παραβίασης των κανόνων μπορούμε να ενσωματώσουμε το σύστημα παρά αν ε, είχαμε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, και οι δύο χώρες που δεν συνεργάζονται και δεν συμμετέχουν σήμερα στην ενισχυμένη συνεργασία κάποια στιγμή ελπίζω να προσχωρήσουν στους 25 και έτσι να έχουμε πλήρη ε, ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και στο θέμα των ευρεσιτεχνιών. Τώρα αξιοποιούμε τις δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας. Ωραίο θα ήταν όμως αν όλοι συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής εξ ονόματος του Συμβουλίου ο κύριος Λούκα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στη θέση να ανακοινώσω ότι κατά τη χθεσινή σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας οι υπουργοί μα ομόφωνα ενέκριναν τη δέσμη για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ η ιδέα ενό ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματο διπλωμάτων ευρεσιτεχνία ανάγεται στη δεκαετία του 1970, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ήδη από τότε ήταν ευρέως παραδεχτό ότι ένα τέτοιο σύστημα θα έδινε σημαντική όθηση στην ανταγωνιστικότητα της καινοτόμου βιομηχανίας μας δημιουργώντας μια ενιαία αγορά ευρεσιτεχνιών. έκτοτε η πορεία υπήρξε μακρά και η πρόοδος κατά καιρού σποραδική. τώρα όμως η κατάληξη είναι πλέον ορατή και θα ήθελα να αρχίσω χαιρετίζοντα το γεγονό ότι είμαστε στα πρόθυρα της θέσπισης ενός ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση του συστήματος αυτού θα δίνει τη δυνατότητα απλής και οικονομικά συμφέρουσας πρόσβασης σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας υψηλής ποιότητας που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα θα προσφέρει προβλέψιμη και αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας η θέσπιση του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας σημαίνει ότι το κόστος της απόκτησης προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση αναμένεται να μειωθεί κατά 80% μπορεί και περισσότερο. Σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει τον μέσο όρο δαπάνης για κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από 36.000 ευρώ σε 4.700 ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μείωση η οποία θα επιτρέψει στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας να διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές ανάλογες εκείνων των ισχυρών στις αγορές των ε, βασικότερων ανταγωνιστών μας της ιαπωνίας και των ηπα θα επιτρέψει επίση τα διπλώματα ευρεσιτεχνία να καταστούν πιο προσιτά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. όμω τα υψηλά ποιότητα και οικονομικώ αποδεκτά δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία πρέπει να συνοδεύονται από ένα σύγχρονο και εναρμονισμένο δικαστικό σύστημα που θα μπορεί να εγγυάται νομική ασφάλεια και δικαστικέ αποφάσει υψηλή ποιότητα σε λογικό κόστο κάτι τέτοιο θα βελτιώσει σημαντικά την εμπιστοσύνη της βιομηχανίας στο σύστημα. για να αξιοποιηθεί στο ακέραιο το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χρειάζεται ειδικευμένο δικαστήριο που θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και θα κατοχυρώνει την νομική ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διαφορών σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση γι' αυτόν τον λόγο τον ερχόμενο φεβρουάριο θα συναυθεί σχέδιο διεθνούς συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη σύσταση ενιαίου ειδικού δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με αποκλειστική δικαιοδοσία έπτων των διαφορών που αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ενιαία ισχύ. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο συμμερίστηκε απολύτως την αποφασιστικότητά μας να υλοποιήσουμε ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνία ποιοτικά υψηλό και προσιτό από το οποίο μπορούν να ωφεληθούν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτιμώ πολύ τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο τα δύο θεσμικά μας όργανα μπόρεσαν να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα ήθελα ιδιαίτερα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς τους κυρίους Ράπχεϊ, παλτασαρέ και λένε για το έργο τους ως εισηγητές των τριών συμπληρωματικών μερών του φαγγέλου αυτού οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο δίνοντας μας την δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαι πεπισμένο ότι η δέσμη που βρίσκεται σήμερα μπροστά μα συνιστά ένα νομικό στιβαρό κείμενο που επιφυλάσσει προεξάρχοντα ρόλο στο δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, προσδοκούμε ότι και τα 27 κράτη θα μπορούσαν να προσυπογράψουν τη δέσμη αυτή. Λυπούμε διότι αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα δίχως τη συμμετοχή όλων. Η επιλογή για ενισχυμένη συνεργασία χρησιμοποιείται πάντα ως ίστατο μέσο όταν όλες οι άλλες επιλογές έχουν αποκλειστεί. Στην παρούσα περίπτωση το δίπλωμα ευρεσιτεχνία έχει τόση σημασία για τη μελλοντική μα ανταγωνιστικότητα που δεν είχαμε την πολυτέλεια να περιμένουμε περισσότερα από ό,τι κάναμε ήδη. ευελπιστώ πάντω ότι και τα εναπομείναντα κράτη μέλη θα μπορέσουν να υιοθετήσουν το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία στο προσεχέ μέλλον. σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Και τώρα ο Επίτροπος Μπαρνιέξ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα αξιότιμου βουλευτέ. βουλευτές. ακούσαμε από τον Υπουργό Μόλι τώρα, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος ενό μακρύτατου δρόμου. Διαδοχικές προεδρίες εργάστηκαν για αυτό το ζήτημα εδώ και δύο χρόνια. Κυρίως η Κυπριακή Προεδρία που δραστηριοποιήθηκε όλος ιδιαίτερος για αυτό το ζήτημα και είστε μάρτυρες ε, αυτού του δρόμου που διανύσαμε. Όπως ε, και οι βουλευτές, ε, θέλω να τονίσω, όπως είπε και ο Πρόεδρος λένε και οι συγητές Ραπκά και Μπαλτασάρε, κατέδειξαν μεγάλη επαγγελματική επάρκεια και υπομονή. Καθώς και μία ένα γνήσιο ενδιαφέρον ε, για την ευρωπαϊκή ιδέα. Μπορούμε με τη βοήθεια της Επιτροπής ε, να ολοκληρώσουμε αυτό το μακρύ, το υπερβολικά μακρύ δρόμο που χρειάστηκε να διανύσουμε τόσο ώστε να κατοχυρώσουμε προστασία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Τη δεκαετία του 60 ξεκίνησε αυτή η συζήτηση σε διάφορες φάσεις με διαδοχικές αποτυχίες και το 2010 είχα εκφράσει ενώπιόν σας ε, την ελπίδα Χωρί να είμαι και ο πρώτο επίτροπος, Ευρωπαϊο επίτροπο ε, που επιλαμβάνεται του ζητήματο, εξέφρασα λοιπόν την επιθυμία μου να είμαι ο τελευταίο. Ε, χάρη στην αποστήριξή σα, ελπίζω να ευοδοθούν οι προσπάθειε μα. Ε, τα στατιστικά στοιχεία που μα έδωσαν οι συγγητές τώρα στη ΣΥΠΑ το 2011, κυρίε και κύριοι, οι Αμερικανοί κατέθεσαν 224.000 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε ένα χρόνο. Στην Κίνα 170.000. 172.000. Αναφερθήκατε και εσείς στην ε, Κίνα, τα δικά μας στοιχεία είναι 62.000 ε, μόνο, είναι ένας από τους λόγους, όχι ο μοναδικός, που εξηγούν την περιπλοκότητα και το κόστος που συνεπάγεται η προστασία των διπλωμάτων ε, στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς. Σήμερα σημειώνεται πρόοδο σε τέσσερα σημεία ταυτόχρονα για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα έχουμε ένα δίπλωμα που θα ισχύει σε 25 κράτη-μέλη και όπως μας είπε ο πρόεδρος Λένε, έχει ανοίξει η πόρτα πλέον και δεν θα υπάρξει καμία διακριτική μεταχείριση εις βάρος των ε, Ιταλικών και Ισπανικών επιχειρήσεων. Εξάλλου η μετάφραση μπορεί να γίνει για εμπορική χρήση στα Ιταλικά και στα Ισπανικά. Και επί τη βάση της προόδου που σημειώνουμε από κοινού, ευελπιστώ ότι η Ισπανική και η Ιταλική κυβέρνηση θα μπορέσουν να προσχωρήσουν ε, στο σύστημα, ούτως ώστε το νέο μέσο αυτό να μπορεί να λειτουργήσει ολόκληρη την εσωτερική αγορά, τουλάχιστον το ελπίζω, πάση ειλικρινή από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η μοναπευθυντική θηρίδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνονται κατά αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών για αυτό. Ο Υπουργός μας έδωσε και τα αριθμητικά στοιχεία ε, το κόστος 6-7 ε, φορές ε, και ε, συνιστά αυτό μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εργαστήρια. Τέλος στις διαπραγματεύσεις ε, οι τελευταίες ε, αναταραχές ε, στο Συμβούλιο στρέφονται γύρω από μια ειδική προστασία ούτως ώστε να διευκολυθούν οι διαδικασίες στα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα. Τέλος, διάδοση των πληροφοριών σε όλες τις γλώσσες. Ε, βασιζόμαστε στο τωρινό γλασικό καθεστώς ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου, αλλά ε, τεχνικές υψηλής ποιότητας μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες μετά την καταγραφή του διπλώματος κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι να φτάσουμε στο σύστημα της αυτόματης μετάφρασης θα καθίσταται δυνατό να γίνεται μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και η Ιταλική και η Ισπανική το τονίζω για τη μέγιστη διανο των ε, τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών των ευρωπαϊκών διπλωμάτων Βρεστιχνίας προς όφελος όλων στην εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι ε, θα αλλάξει άρδινη κατάσταση καθότι καταφέραμε πλέον να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση ε, δεν χρειάζεται να ε, προσφύγουμε στην ενισχυμένη συνεργασία, κάτι που επιτρέπει η Ρίστον παρόδο η συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζω λοιπόν να ε, ακολουθήσουν το άρμα της πρόοδου και οι δύο εναπομείνωσες χώρες και αυτές οι τελευταίες αναταραχές, όπως μας είπαν και οι συγητές στο Συμβούλιο, μας θορύβησαν, αλλά πιστεύω ότι καταλήξαμε στη βέλτιστη δυνατή πολιτική συμβαστική λύση για την οικονομία και για τις επιχειρήσεις. Τέλος, ε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι με την έγκριση αυτού του σχεδίου ε, βάζεται άλλο ένα λιθαράκι σε αυτό το θεματολόγιο που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οικονομία, ε, ανάκαμψη, ανάπτυξη, στα πλαίσια του νομοθετήματος για την ενιαία αγορά 1 και 2 καταθέσαμε περίπου 55 ε, νομοθετικές προτάσεις ε, συγκεκριμένες που διευκολύνουν τις διαδικασίες, ε, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πολιτών, επαγγελματικές δεξιότητες παραδείγματος χάρη, τα μέτρα για τη διαφάνεια ως προς τις τραπεζικές δραστηριότητες, κοινωνική επιχειρηματικότητα, ηλεκτρονικές υπόψεις, υπογραφές, ε, ψηφιακό θεματολόγιο, ε, διπλώμα ευρεσιτεχνίας. Είναι μάλλον η πιο συμβολική κίνηση από όλες. Ε, βρίσκονται επιτάπητος όλες αυτές οι προτάσεις θα εξεταστούν από το Κοινοβούλιο και τους Υπουργούς. Η οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες χρειάζονται αυτά τα μέτρα. Πρέπει να περάσουμε συγκεκριμένα μηνύματα ότι εργαζόμαστε υπέρ της προόδου των Ευρωπαίων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας Ενέργειας, ο κύριος Μετσάρος, δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους δύο τους συνεισήγητες για τη συνεργασία τους και την εξαιρετική δουλειά την οποία τελικά έκαναν σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια καινοτόμο κοινωνία. Φυσικά να προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία. Το νέο σύστημα, το ενιαίο αυτό σύστημα, είναι κάτι το οποίο θα υπηρετήσει τους προηγούμενους στόχους. Αναζητούσαμε ένα νομικό ενιαίο πλαίσιο για δεκαετίες το οποίο κυρίως να προστατεύει και να απλοποιεί το σύστημα. Βλέπουμε ότι υπήρχαν εμπόδια μέχρι τώρα στην βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει αρχίσει και μένει πίσω στον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε λοιπόν τώρα σε θέση να δώσουμε περισσότερες εγγυήσει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος βέβαια το οποίο θα μειωθεί στα πλαίσια της κατάθεσης των νέων αιτήσεων, αλλά στην ουσία θα βοηθήσουμε και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Θα καταστήσουμε την Ευρώπη περισσότερο ανταγωνιστική, θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή σκηνή. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν και το, την λεγόμενη μονοαπευθυντική θηρίδα, και οι διαδικασίες θα απλουστευθούν και δεν θα υπάρχει αυτό το παλαιό σύστημα που έπρεπε κανείς να περνά από όλε ε, τις χώρες. Ε, λυπάμαι που κάποιες χώρες σε αυτή τη φάση δεν συμμετέχουν, ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα αναθεωρήσουν την άποψή τους. Η δημιουργία ομοιομορφία στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δημιουργήσει ασφάλεια και σταθερότητα. Είναι ένα σύστημα ευεργετικό για τις μικρομεσαίες, όπως επίσης ε, και τις ε, νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται, τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις λεγόμενες startup. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Επόμενη ομιλήτρια για τέσσερα λεπτά η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Επίτροπε, αξιότιμε Υπουργέ Λουκά, αξιότιμοι εισηγητές. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την ε, συμφωνία που υλοποιεί τον στόχο του Ευρωπαϊκού Συστήματος με ενιαίο σύστημα μετά από 50 χρόνια. Πριν από το καλοκαίρι θεωρούσαμε ότι θα είχε εξευρεθεί συμβιβαστική λύση και θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Μετά το Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο μας διεμήνησε τη διαγραφή τριών παραγράφων πράγμα που απογοήτευσε και φόβησε το Κοινοβούλιο. Πολλές φορές ε, είχαμε παρόμοιες εξελίξεις, ποτέ όμως τόσο μη παραβίαση των ε, κανόνων μας. Ε, μη νομοθετικό όργανο παρενέβη ε, και εξευρέθη συμβιβαστική λύση που άλλαξε την καρδιά του νομοθετήματος και κατέστη ε, νομοθέτημα που παραβιάζει τις συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας χάρη στους τρεις εισηγητές που πίεσαν ε, πεισματικά ε, για την αποκατάσταση των άρθρων ε, μπορέσαμε να βρούμε μια λύση. Δεν είναι ιδεώδης, αλλά το Κοινοβούλιο εξασφάλισε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει την αρμοδιότητα και θα είναι το μόνο το οποίο ε, ερμηνεύει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Συνταγματικής Επιτροπής θα ήθελα να τονίσω ότι ε, μια πιο αποτελεσματική προστασία θα ωφελήσει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν την κρίση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ε, η ε, ε, επικύρωση μπορεί να γίνεται στα κράτη-μέλη και θα είναι αρμόδιο το δικαστήριο σε περίπτωση διαφοράς. Ε, μόνο με αποτελεσματικό σύστημα μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο υπέρτατος στόχος είναι να τηρείται το ενωσιακό δίκαιο και το δρόμος προς το δικαστήριο μέσω προδικαστικών αποφάσεων με βάση το αντίστοιχο άρθρο θα είναι δρόμος ανοιχτός. Και αυτό μπορούσε να το διασφαλίσει το Κοινοβούλιο. Απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη όλα να συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία ε, και να δημιουργήσουν διεθνή συμφωνία ε, για τις, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ε, θα πρέπει να ε, υπάρχει γνήσια ενισχυμένη συνεργασία από όλους. Τέλος θέλω να τονίσω και να θυμίσω πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη ε, να προωθήσουμε τους καινοτόμους ανθρώπους και να εγγυηθούμε για τις εφευρέσεις τους με το λιγότερο δυνατό κόστος και γραφειοκρατία για να επιβιώσουν και οι μικροί δεν, θα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής προστασία αλλά και επαρκής προώθηση, ενίσχυση των ευρεσιτεχνών με τις αντίστοιχες πιστώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε και τώρα οι αγορητές εξ των πολιτικών ομάδων. Εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τέσσερα λεπτά ο κύριος Σφίφκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα μετά από τους πολλούς μήνες σκληρή εργασία για την συγκρότηση του ενίου συστήματος προστασίας και κατοχήρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εσωτερική αγορά να έχουν τη θέση που του αναλογεί στην ε, διεθνή οικονομία. Μεσούσει της ε, κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του να είμαστε να έχουμε μια εξελιγμένη οικονομία ώστε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ε, απασχόλησης, θα πρέπει να ε, βρούμε λύσεις για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σήμερα νομικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Είναι θεμελιώδης σημασίας ε, η πρόοδος που σημειώνουμε σήμερα, διότι όπως είπα θα επιτύχουμε τους στόχους μας, θα, αναγκαστικά θα γίνουμε πιο καινοτόμοι Ε, το υψηλό κόστος ε, που συνδέεται με την κατοχήρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, παραμένει δυστυχώς. Υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες που θα βοηθούσαν στην παγκόσμια εμπορική σκηνή να ενισχύσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μένουν ε, σκονισμένες ε, μέσα στα συρτάρια αυτές οι ενδιαφέρουσες ε, ιδέες. Ερευνητές στην Πολωνία μου είπαν, Φερρυπίν, ότι δεν ωφελεί το δίπλωμα έβρεση τεχνίας λόγω του υψηλού κόστους και αυτό που θα αποκόμιζαν από την χρήση της τεχνίας στη βιομηχανία είναι αμεληταίο σε σχέση με το υψηλό αυτό κόστος. Ελπίζω λοιπόν να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εγώ ε, θα ήθελα να είχαμε ολοκληρώσει νωρίτερα ε, αυτό το έργο, αλλά δεν συνέβη. Αλλά τι να πει κανεί, μια μικρή καθυστέρηση μπροστά σε δεκαετίες διαπραγματεύσεων ε, δεν είναι τόσο σημαντικό όταν θυμάμαι ε, τον ενθουσιασμό που μας χαρακτήριζε επί Πολωνικής Προεδρίας όταν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, λυπάμαι διότι λόγω της ε, ανάρμοστης συμπεριφοράς του Συμβουλίου και λόγω ε, των παρανοήσεων που δημιουργήθηκαν μετά από κάποιες αντιπαραθέσεις, μόνο τότε μπορέσαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα τον κύριο Κάμερον και τους Βρετανούς συναδέλφου μας για τι ιδέε που κατέθεσαν ώστε να αλλάξει η κατάσταση. αναβαθμίζοντας την προστασία των Βρετανικών ε, κυρίως ε, συμφερόντων. Χαίρομαι για την ευτυχή κατάληξη, αλλά ας μην είμαστε συγκαταβατικοί και αυτάρεσκοι. Η θέσπιση ενός ε, συστήματος ενιαίας ε, προστασίας και ενός ειδικού δικαστηρίου είναι στοιχεία κλειδιά ναι μεν, όμως θα πρέπει να μεριμνήσουμε ταυτόχρονα να είναι συνετή και λογική η διαδικασία ε, κατοχύρωσης για τις βιολογικές διεργασίες παραδείγματος χάρη ή για τις εφευρέσεις ή λογισμικά Φετρές που σχετίζονται με την πληροφορική και τα λογισμικά. Ε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε περισσότερους ανταγωνιστές από ό,τι υποστηρικτές. Να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και χαίρομαι πολύ που παρατώθηκε επιτέλους αυτή η μακρόχρονη διαδικασία. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κ. Κοφεράτη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε αγαπητοί συναδέλφοι. Έχουμε καταλήξει ένα βήμα πριν από το τελικό αποτέλεσμα, το τόσο σημαντικό. Το αποτέλεσμα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους τον τελευταίο μήνα ε, που θα οδηγούσαν σε μια αποτυχία της ε, πρώτης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, να προωθήσει ένα θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση από το 1957 και μας επέτρεψε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ορισμένα σημαντικά νομικά εμπόδια. Η προστασία του συστήματος ευαισθητεχνίας στο εσωτερικό της Ένωσης είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την ανάπτυξη της Ευρώπης και για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό δείχνει επίσης και τη μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου κατάφερε να προωθήσει μέτρα πολύ σημαντικά για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υποστηρίξει επίσης τις επιχειρήσεις αυτές το κόστος των μεταφράσεων στις γλώσσες πέραν της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής πέρα από το θέμα το γλωσσικό το οποίο έγινε αντικείμενο καταχρηστικών ερμήνειων θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα το οποίο προωθεί το πακέτο το οποίο έχουμε μπροστά μας δεν αποκρύβει θα έλεγα τα μέτρα τα οποία προστατεύουν τις επιχειρήσεις οι οποίες γλωσσικά δεν εκπροσωπούνται σε αυτό το τριπλό γλωσσικό σύστημα. Την του Συμβουλίου του Ιουλίου το Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει να αναβάλει την ψηφοφορία στο πακέτο των προτάσεων και είχε εκφράσει την αγανάκτησή του απέναντι στην απαράδεκτη στάση του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα πήρε δύο πολιτικές αποφάσεις, το να μην μετατρέψει το θέμα σε μια διοργανική μάχη και να καταλήξει σε μια λύση συμβατή με τις συνθήκες μετά από αντιπαραθέσεις πέντε μηνών καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία ικανοποιεί θα έλεγα τις απαιτήσει που θέτει η νομική βάση στα πλαίσια της ενιαίας προστασίας και σεβόμενη και τον σεβασμό επίσης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η εμπλοκή στην ομοθετική διαδικασία του Συμβουλίου είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι καταλήξαμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα που σέβεται τους στόχους που είχαμε θέσει, λιγότερο κόστος, μεγαλύτερη προστασία, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη νομική διασφάλιση. Έχουμε ανάγκη από ένα τέτοιο σύστημα κάτι το οποίο θα βοηθήσει το σύνολο του οικονομικού μας συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, η κυρία Βίξτρομ για τρία λεπτά. Ουσιαστικά υπάρχει μία λέξη που δημιουργεί αυτή τη συγκίνηση. Επιτέλους. Επιτέλους καταφέραμε να φτιάξουμε στην, αυτό που απέτυχε να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρότι γνώριζαν όλοι πόσο θετικό θα ήταν αυτό για τους εφευρέτες, ε, για, τους, ε, για τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και ούτω καθεξής. Ήταν μακρύς και δύσκολος ο δρόμος και τελικά χρειάστηκε μια ενισχυμένη συνεργασία 25 κρατών από τα 27 για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα ήθελα όμως σήμερα να τονίσω επίσης ότι η πόρτα για την ε, Ιταλία και την Ισπανία προς το παρόν απέχουν είναι ορθάνυχτη και καλωσορίζουμε αυτές τις χώρες με το που το θελήσουν μπορούν να προσχωρήσουν στο σύστημα και ελπίζω να προκρίνουν τον κοινό δρόμο στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερο τον Επίτροπο Μπαρνιέ για τη δική του συμβολή και την απίστευτη εργασία ολόκληρου του επιτελείου του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάρη στον Επίτροπο ε, μπορέσαμε τελικά να επιτύχουμε το στόχο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Λένε Ραπκάη και Μπάλτασάρε, τους τρεις εισηγητές του Κοινοβουλίου με την, το επικοδομητικό τους έργο μας οδήγησαν ε, στην ευτυχή κατάληξη αυτής της διαδικασίας. Από πλευράς των φιλελεύθερων ανέκαθεν ήταν ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ταυτόχρονα θα έχουμε ένα ειδικό δικαστήριο για την ρύθμιση των διαφορών και στο μέλλον δεν θα έχουμε δεκαπλάσιο κόστος για την κατοχήρωση σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα η επιχείρηση δεν χρειάζεται να εμπλέκεται σε παράλληλες πολλές ε, δικαστικές ε, διαδικασίες σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ενιαία προστασία με ένα μόνο αρμόδιο δικαστήριο και μια ενιαία δικαιοδοτική διαδικασία. Έτσι θα επιτύχουμε την ισορροπία στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα κατοχήρωσης της ευρεσιτεχνίας και θα απαλείψουμε τα περιτά γραφειοκρατικά άχθη. Είναι μια ιστορική ημέρα η σημερινή και πρόκειται για ένα ορόσημο στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ευημερία και ανάπτυξη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μόνο έτσι θα εξέλθουμε από την κρίση στην Ευρώπη. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι πανάκια το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι όμως ένα από τα μέσα που θα την ανάπτυξη και την ευημερία στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενη ομιλήτρια εξ ονόματο τη Ομάδα των Πρασίνων για 3,5 λεπτά η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ευρεσιτεχνιών, ευρωπαϊκό σε εισαγωγικά. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, αποφασίζει σε σχέση με τη νομική βάση. Αυτό πάντα ήταν κάτι που το σεβόμεθα. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Διευκρινίζω. Πάντοτε έδινα μάχη για ε, ευρωπαϊκό σύστημα ευρεσιτεχνιών, το οποίο θα ήταν προσιτό, που θα μπορούσε να ωφελήσει τους χρήστες, θα ήταν οικονομικό και θα μπορούσε να μας πάει μπροστά δεν πληρούνται σήμερα οι προϋποθέσεις αυτές. Ο συνόδελφος Κάι αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης αυτής που ήταν πολύ προβληματική αναμφίβολα. Εκεί που διαφέρομαι είναι η κρίση μας σε σχέση με τη συμβιβαστική λύση που έχουμε μπροστά μας αφότου το Συμβούλιο έβγαλε τα κεντρικά άρθρα αυτής της ρύθμισης μετά από επιθυμία του Κάμερον για να τα λέμε σωστά. Η συμβιβαστική αυτή λύση που εξευρέθη πλέον με διεθνή συμφωνία δεν είναι αυτό που θα δημιουργήσει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Να το πούμε καθαρά. Εμείς τις δυνατότητες μας άσκησης επιρροής δεν τις ασκούμε, παρετούμεθα από αυτές. Μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ελάχιστες δυνατότητες προβλέπει για ένσταση, ξέρετε, την διαδικασία των προδικαστικών αποφάσεων. Ε, πάντοτε θα πρέπει να θέτουμε και το επόμενο ερώτημα εδώ. Ποιον ωφελεί λοιπόν η ρύθμιση αυτή, το σύστημα γίνεται ακόμα συνθετότερο. Αυτό που είναι σύνθετο προκαλεί δυσκολίες στις μικρομεσές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν ωραιότατα να, να πάρουν ολόκληρη στρατιά από δικηγόρους και να βγάλουν υπέρ αυτών αποφάσεις. Για τις μικρομεσαίες είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό ήρθαν σε εμά και μας είπαν παρακαλώ όχι έτσι, δεν θα μας βοηθήσει αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δεύτερο σημείο μεγάλες ε, επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών ενίστανται εντωμεταξύ και λένε ότι δεν θέλουμε αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το θέμα του κόστους. Μάλιστα, το μπορεί να φτηνίνει ε, το δίπλωμα να το πάρει κανείς αλλά τα δικαστικά έξοδα λόγω της αυξημένης συνθετότητας του προβλήματος θα αυξηθούν και αυτό θα βλάψει ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες. Η επιστημονική κοινότητα το απορρίπτει το μοντέλο και τη συμβιβαστική λύση ε, η οποία στη γνωμοδότηση προδικάζεται. Ε, τώρα, ε, λίγα λόγια ακόμα για την πράξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εύρεση Τεχνίας που πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια του τι είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί με δίπλωμα εύρεση τεχνίας είτε πρόκειται για εφεύρεση, για προνόμια ή το λογισμικό που θα πρέπει να συνοδεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έχουμε πολύ μειωμένε δυνατότητες να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να διασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως το είχαμε φανταστεί και γι' αυτό δεν μπορώ να συγκατατεθώ σε αυτό. Δια... Διακινδυνεύει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να προστατεύει. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ε, για δύο λεπτά ο κύριος Καρύμ για τους Ευρωπαίους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ηγητέ και τον Επίτροπο Μπαρνιέ, διότι αναγνωρίζεται ο ηγετικό του ρόλο και τον καλωσορίζουμε. Συνάδελφοι, ειδού το ιδανικό παράδειγμα τη δυσλειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρονολογικά, αν εξετάσουμε το ζήτημα, θυμάστε πριν από λίγα χρόνια ότι όλοι ζητούσαν αυτά τα μέτρα. Και εμείς τι απάντηση δώσαμε, περιμένετε τέσσερις δεκαετίες και βλέπουμε στην Επιτροπή όταν συζητήθηκε ε, το ενδεχόμενο μια συμβαστική λύση να έχουμε στο Λονδίνο ένα δικαστήριο που ε, επίσημη γλώσσα έχει τα γερμανικά και αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα για άλλε τρει πρωτεύουσε. Ε, καταλαβαίνετε αυτό δεν δείχνει σοβαρότητα για την λύση που τελικά επιλέξαμε. Πάντω χρειαζόμαστε αυτό το μέτρο και πρέπει να επισπεύσουμε τι κινήσει μα όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα αλλά και σε άλλα. Η Κίνα, νιώθουμε την ανάσα θα της Κίνας ε, ε, δίπλα μας ε, και όσοι ασχολούνται με τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Ινδία θα έπρεπε να μιλήσει με τους συνομιλητές για την ενίσχυση των διατάξεων για τη δική τους προστασία. Όταν κάνω μια αντιπαραβολή ανάμεσα στο δικό του σύστημα και το δικό μας, τους ζηλεύω. Είμαστε πλέον ουραγοί. Να σας πω τι γίνεται στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή. Έχουν εκδώσει τρεις φορές περισσότερα διπλώματα σε σχέση με εμά και διπλάσιος είναι ο αριθμός ε, όταν βλέπουμε τι συμβαίνει στην Κίνα. Ε, η Κίνα, η Ιαπωνία και η ΙΠΑ από κοινού εκπροσωπούν το 82% της αύξησης του αριθμού των διπλωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπερβάλλουμε όταν ισχυριζόμαστε ότι είναι ζωτική σημασία στο μέτρο και πρέπει να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση. Είναι κατεπήγοντο το ζήτημα και χρειάζεται ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ. Επόμενο ο για 1,5 λεπτό, ο κύριος Μαστάλκα από την ε, ομάδα τη αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ε, πω πόσο ευγνώμων είμαι για τους ασύγητες. Ε, κάνα μια τεράστια προσπάθεια σε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τον χώρο αυτό από τη δεκαετία του τα προβλήματα είναι πολλά και το γλωσσικό και τα θέματα της νομικής αμφισβήτησης και τελικά συμφωνούν οι 25 χώρες με την δεδομένη συμβιβαστική λύση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι χώρες της Ένωσης δεν θα είναι 100% ικανοποιημένες. Αυτή είναι η έννοια του συμβιβασμού. Όμως προχωράμε σε μια απλούστευση της διαδικασίας. Το θέμα είναι όταν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι κανόνες να βοηθήσουν να εξοικονομηθούν χρήματα και να διευκολυνθούν οι πρακτικές διαδικασίες. Ευχαριστώ και την Κυπριακή Προεδρία για την προσπάθεια την οποία κάνει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές το ταχύτερο δυνατόν, περιμένοντας βέβαια και την απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενο ο μιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Πάτεν από την Ευρώπη Δημοκρατίας και Ελευθερίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι μια επιπλέον άχρηστη και μία απαραίτητη μεταφορά αρμοδιότητας από το εθνικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς ε, έχουμε ένα σύστημα το οποίο παράγει στο Ηνωμένο Βασίλειο 750 εκατομμύρια στερλίνες τον χρόνο και τίθεται εν κινδύνο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και για τον διορισμό των μελών στο νέο δικαστήριο και για την ποιότητα των αποφάσεων οι οποίες θα ληφθούν. Στην ουσία ε, υποτίθεται ότι όλες ε, οι χώρες θα έχουν δικαίωμα σε ένα δικαστή ενώ υπάρχουν μικρές χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη εμπειρία και δεν έχουν και εμπειροδικαστικό προσωπικό γύρω από το θέμα της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στην ουσία θα διευκολυνθούν για μια ακόμη φορά οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εις βάρος των μικρομεσαίων. Ε, πάλι το κόστος θα είναι ανυπόφορο για τις μικρές επιχειρήσεις και θα πρέπει να τρέχουν στη Γαλλία, στη Γερμανία για να προστατεύουν τα έργο τους και όχι στα τοπικά δικαστήρια. Οι εμπειρογνώμονες δεν πιστεύουν ότι θα γλιτώσουμε χρήματα. Το κόστος ε, της αμφισβήτησης ε, της εγκυρότητας κάποιων ε, τέτοιων διπλωμάτων θα αυξηθεί, θα τριπλασιαστεί μάλιστα. Κύριε Μπάτεν, μπλε, μπλε κάρτα από τον κύριο Καρύμ. Δέχεστε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Μπάτεν, αυτό το οποίο μας είπατε είναι πραγματικά ανόητο. Αυτό το μέτρο το ετοιμάζουμε εδώ και 40 χρόνια. Πότε εσείς ήρθατε σε μια συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να θέσετε τις αντιρρήσεις σας. Αλλά το κόμμα σας ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα γύρω από το θέμα αυτό και αυτά τα οποία είπατε τώρα είναι απλά μια μεγάλη ανοησία. Ο κύριος Μπάτεν απαντά, ανταπαντά. Ξέρετε ότι δεν είμαι φανατικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παίρνω τις πληροφορίες μου από τον δόκτωρα Γιάκεν Μπάτενμπεργκ, ο οποίος είναι εμπειρογνώμων. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Μονάχου, των Παρισίων ήταν μέλος του πάνελ των εμπειρογνωμόνων και αποχώρησε από το σώμα αυτό το 2011. Λοιπόν, αντίθετα με σας, εγώ δεν είμαι φανατικός αυτού του σώματος και παρόλα αυτά παραπέμπω σε ένα εμπειρογνώμονα ο οποίος γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Πραγματικά ε, κύριε Κάμελ θα ήταν διασκεδαστικό να σας ξαναδώσω για μια ακόμη φορά το λόγο αλλά ε, Λυπάμαι πρέπει να συνεχίσουμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σίλστρα για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το ενίο δίπλωμα είναι εξαιρετική ιδέα. Αυτοματική αυτοματική προστασία, τυποποίηση του κόστους, αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Η ιδέα υπάρχει. Αλλά η πρακτική υλοποίηση είναι τόσο περίπλοκη ώστε η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας γίνεται αβέβαιη. Έχουμε ένα νομικά βέβαιο σύστημα με πολλούς τύπους προστασίας ε, κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περίοδου που και αυτή είναι αβέβαιη. Ε, δημιουργούμε ανασφάλεια ε, αβεβαιότητα, όχι προστασία. Ούτε θα είναι φθηνότερο το σύστημα για τους εφευρέτες, για τις μικρές, τις καινούριε επιχειρήσεις. Ε, το, το κόστος τους θα αυξηθεί και τα, οι νέες ε, έδρες στο Παρίσι, Λονδίνο δεν θα στοιχήσουν φθηνά. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα αν η Ιταλία και η Ισπανία είχαν συμμετάσχει για τα, ως ανταλλαγή για τα εκατομμύρια ε, ευρώ που στέλνουμε προς την κατεύθυνσή τους δεν θα ήταν υπερβολικό να το περιμένουμε από αυτές τις χώρες αυτό. Όμως η Ένωση δεν είναι γνήσια Ένωση. Οι χώρες δεν φαίνεται να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται ούτε οι πολίτες ούτε και οι επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτή η Ένωση είναι μόνο για τους αξιωματούχους και τους πολιτικούς. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για τέσσερα λεπτά, ο κύριος Λόπες Ιστούρες White. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για πάρα πολλά χρόνια παρακολουθήσαμε να λειτουργεί ένα σύστημα, προσπαθήσαμε να πετύχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ενιαίο που να ισχύει στο σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους. Εγώ στηρίζω τις προτάσεις αυτής έτσι ώστε να ενταχθεί στο κοινοτικό δίκαιο το σύστημα χορήγησης διπλωμάτων ένα σύστημα το οποίο δεν πρέπει να προκαλεί διακρίσεις, να σέβεται τις αρχές της συνθήκης σε σχέση με την εδαφική και κοινωνική και οικονομική συνοχή, να δημιουργεί ένα αίσθημα νομικής διασφάλισης και βεβαιότητας και να κινητοποιεί την καινοτομία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις βασικές αρχές τις συμμεριζόμεθα όλοι βέβαια. Πάντως ε, ε, το σύστημα έτσι όπως παρουσιάζεται έτσι όπως έχει σήμερα δεν δημιουργεί νομική βεβαιότητα, προκαλεί υπερβολικά κόστη και δεν προωθεί την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η άποψή της ήταν η καλύτερη, θέλησε να την επιβάλλει και γι' αυτό έτσι κι αλλιώς η δυνατότητα που δίνεται για τη νομική αμφισβήτηση σε ένα δικαστήριο με τρεις έδρες το οποίο δεν είναι καθόλου ενιοποιημένο στην ουσία ε, είναι μια προέκταση της λογικής της διακυβερνητικής συνεργασίας. και είναι κάτι το οποίο παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει ο στόχος είναι ευγενής και θετικός, καλός, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε χώρες όπως η δική μου όπου το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να παίρνουμε μέτρα τα οποία θα είναι αντίθετα με την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Ο κάτοχος του τεχνίας θα έχει ε, δυνατότητες και δικαιοδοσία θα έλεγα αποκλειστική και μονοπωλιακή σε σχέση με τη χρήση ενώ θα έπρεπε να προστατεύσουμε φυσικά τους εφευρέτες αλλά ταυτόχρονα να προωθήσουμε και την εμπορική δραστηριότητα και εκμετάλλευση. Έχουμε λοιπόν κάνει μέτρα, έχουμε προτείνει μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν είναι ικανοποιητικά. Για μία ακόμη φορά περνάμε σε πολυδιάσπαση της εσωτερικής αγοράς και ε, θα πρέπει να περιμένουμε και οι 25 χώρες να δημιουργήσουν το ενιαίο αυτό δικαστικό σύστημα. Είναι περίπλοκο το σύστημα αυτό και ο μεγάλος αριθμός των δικαστηρίων για την επίλυση των διαφορών είναι ένα σύστημα το οποίο θα κοστίζει πάρα πολύ είναι ένα σύστημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί την επιθυμητή νομική ασφάλεια και το σύστημα και οι ρυθμίσεις που προτείνονται για τη γλωσσική πλευρά, για τις μεταφράσεις δεν είναι ικανοποιητικοί. Κάποιες χώρες θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους, κάποιες άλλες χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες, κάτι το οποίο θα δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια σε επίπεδο ε, των εφευρέσεων των διπλωμάτων ευαισθητεχνίας πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα σε όλες τις γλώσσες και όχι μόνο σε τρεις, σε όλα τα δικαστήρια και όχι μόνο σε τρία. Νομίζω ότι τα θεμέλια αυτής της προσπάθειας είναι ιδιαίτερως ασθενή. Είναι κάτι το οποίο είναι θα έλεγα θετικό μόνο θεωρητικά όπως έλεγαν οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Max Planck, χάσαμε την δυνατότητα με τις παρούσες προτάσεις για να εξυγχρονίσουμε πραγματικά το σύστημα. Μόνο αν σεβαστούμε το πνεύμα και το γράμμα των συνθήκων θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση η οποία να ισχύει και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Επόμενη ομιλήτρια για δύο λεπτά η κυρία Γκέρνιερ Ντεόντεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από 30 χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων επιτέλους μπήκαμε στην τελική ευθεία και έχουμε το συμβιβαστικό πακέτο επιτάπητος ε, που θα μπορέσει να προστατεύει τις εφευρέσεις μας σε 25 κράτη-μέλη. Το σύστημα θα απλουστευθεί πολύ σε σύγκριση με το παρόν και το κόστος θα μειωθεί κατά 80%. Επιτέλους λοιπόν θα έχουμε ένα μέσο για την προστασία της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος των διπλωμάτων είναι δεκαπλάσιο από ό,τι είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το συνολικό κόστος ε, είναι περίπου 25.000. Χάρη στην πρόταση αυτή θα περικοπεί πέντε φορές πολλές εφευρέσεις ε, πολλούντος εκείνων που προσέφερε την υψηλότερη τιμή από ε, την άλλη ε, όχθη του Ατλαντικού γιατί πολλές φορές οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν για το δίπλωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει νέο σύστημα, προτείνει ένα μέσο ασφαλέστερο και οικονομικότερο. Κάθε επιχείρηση θα μπορεί τώρα να αποφασίζει η ίδια για το τι είναι καλύτερο για εκείνη. Αν θα υπάρχει το εθνικό δίπλωμα, το ευρωπαϊκό, το οποίο θα ισχύει σε μία ή περισσότερα κράτη-μέλη ή το ενιαίο δίπλωμα που συζητούμε τώρα. Πρόκειται για μια ευκαιρία για όλους, ακόμα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι ε, υπάρχουν στοιχεία που τις διευκολύνουν και θα υπάρχει και πρόσθετη χρηματοδότηση για τη μετάφραση για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητική η συμβιβαστική λύση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα επίμαχα άρθρα 6 με 8 έχουν ε, περάσει σε διοργανική συμφωνία και τώρα έχουμε σωστή την κατάλληλη νομική βάση και ένα πολύ λειτουργικό κείμενο. Έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο δεν τροποποιήθηκε πολύ σε σύγκριση με το αρχικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τον Επιτρόπο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενος ομιλη... Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Τάιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Υπουργέ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό οι επιχειρήσεις μας περίμεναν αυτή τη μέρα, κυρίως οι μικρομεσαίες. Εδώ και δεκαετίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε για ενιαία προστασία των διπλωμάτων. Τώρα η απονομή ενός διπλώματος αναγνωρίζεται σε κάθε κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να γίνει αίτηση χωριστά σε κάθε ένα. Αυτό ε, είναι καθαρή γραφειοκρατία που δεν ανταποκρίνεται σε επιταγές των καιρών και από την άλλη αυξάνει πάρα πολύ το κόστος η ευρωπαϊκή προστασία αυξήσει, ε, στοιχίζει το τετραπλάσιο από ό,τι στις είπα. Η Κίνα μας κοροϊδεύει εδώ και καιρό διότι ε, ζητάμε διπλώματα από εκείνους αλλά δεν έχουμε σωστά εδώ. Ε, το, το, τα οφείλουμε όλα αυτά που αποφασίζουμε σήμερα και στους, στις επιχειρήσεις και στους ε, εφευρέτες. Ε, οι μεταφράσεις ήταν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Τώρα όμως εντωμεταξύ έχουμε και την αυτόματη μετάφραση ε, που τελειοποιείται, βελτιώνεται και ούτως ή άλλως ε, τα περισσότερα διπλώματα απονέμονται στα αγγλικά σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα ε, στις αναφορές που πήραμε στη Γερμανία. Δεν, αναφε... δεν ισχύει ότι υπονομεύεται το μονοπόλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οτιδήποτε άλλο δεν θα συνείδε με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ούτε ισχύει ότι εδώ ε, μιλάμε για αποφάσεις σχετικά με τα διπλώματα στο λογισμικό. Ε, οτιδήποτε άλλο επίσης δεν αλλάζει σε όλα αυτά η νομική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Τρία λεπτά τώρα ο κύριος Έγκστρομ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πράσινοι και το κόμμα των πειρατών επιθυμούσαν σύστημα νέας προστασίας και νέο δίπλωμα και ακόμη το επιθυμούμε. Αν αυτό σήμαινε ότι θα είχε ενταχθεί στις πολιτικές και νομικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώ. η πρόταση αυτή, και φαίνεται ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ αυτής, αντιβαίνει σε αυτούς τους στόχους. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απεμπολεί όλες τις πολιτικές αρμοδιότητες για το μελλοντικό σύστημα ε, προς όφελος μιας διακρατικής συνεργασίας ε, που εκπίπτει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το νομικό σύστημα που θα διέπει το ενιαίο δίπλωμα θα εκπίπτει, ξαναλέω, του ε, ένομου συστήματο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κακό για την καινοτομία και για πολλού άλλου τομεί στην Ευρώπη. Γιατί αυτό έχει σημασία, θα σα εξηγήσω. Εδώ και δεκαετίε, όπως ακούσαμε, Λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Είναι ένα διεθνή οργανισμό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό ελέγχου τη Ένωση και εκτό ελέγχου του Κοινοβουλίου. Και είδαμε σε τι μα οδήγησε αυτό. Η συνθήκη που είναι η βάση της λειτουργίας ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών ε, προβλέπει ξεκάθαρα ότι για τα λογισμικά, για ζωντανούς οργανισμούς κτλ. δεν προβλέπεται κατοχήρωση. Όμως το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, χορηγεί ούτως ή άλλως τα διπλώματα. Δεν το λαμβάνει υπόψη. Για τα λογισμικά, παραδείγματος χάρη λένε όχι, όχι, ε, ε, ε, αυτές, αυτά καθε αυτά τα διπλώματα απαγορεύονται, αλλά προβλέπονται όμως για τα λογισμικά τα οποία είναι εν λειτουργία μέσα σε έναν υπολογιστή. Ε, μα αυτά είναι ανοησίες. Θα έπρεπε το σύστημα να υπάγεται σε πολιτικό και νομικό έλεγχο. Χάσαμε όμως αυτή την ευκαιρία και όλη την εξουσία την μετακυλήσαμε σε αυτή τη διακρατική οργάνωση που δεν εμπίπτει στο δίκαιο της Ένωσης. Απευθύνω θερμή έκκληση προς συναδέλφους να επανεξετάσουν το θέμα γιατί είναι εντάξει υπάρχει διάσταση απόψεων για το ζήτημα αλλά υπάρχει κάτι επί το οποίο συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλό για την οικονομία και την καινοτομία κάτι στο οποίο αποσκοπούμε. Ενώ ένα ε, σύστημα που δυσλειτουργεί είναι επιβλαβές και επιζήμιο. Δεν έχει νόημα να απεγγυθούμε των δικαιωμάτων μας και να μην κάνουμε αυτό που προβλέπεται να κάνουμε βάσει της νομοθεσίας. Υποστηρίξτε τις τροπολογίες μας, ε, σας παρακαλούμε, ώστε να ανοίξει ο δρόμος ε, για τη θέσπιση ενός πραγματικού ενιαίου συστήματος. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Για ένα λεπτό, ο κύριος Κοσούσνικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συναδέλφοι. Είπε ο Επίτροπος Μπαρνιέ πως ε, επιθυμεί να είναι ο τελευταίος Επίτροπος που ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Τον γνωρίζω, γνωρίζω με ποιο τρόπο εργάζεται και το εύχομαι καλή τύχη. Και καλή τύχη εύχομαι και στον κύριο Ραπκάη, καθώς και σε, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ένωσης. Είναι το πακέτο που εγκρίνεται είναι καλό για τη μείωση του κόστος, αλλά και πάλι θα υπερβαίνει το κόστος σε σχέση με το κόστος της ΕΥΠΑ ε, κατά 800 ευρώ. Ε, και δεν ξέρω αν θα επιτύχουμε την, ε, το στόχο μας για τη διανομή των επιστημονικών πληροφοριών στην ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα και επιχειρηματική κοινότητα. Χρειαζόμαστε μια καλή αυτόματη μετάφραση και ένα ισχυρό σύστημα πληροφορικής ε, για να επιτύχουμε τα αναμενόμενα οικονομικά ωφέλη Ελπίζω λοιπόν να πιστούν οι χώρες που δεν συμμετέχουν μέχρι στιγμής με τη λειτουργία του νέου συστήματος και τελικά να προσχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Σενίν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πακέτο το οποίο μας προτείνεται υποτίθεται για λόγους ορθολογισμού και οικονομίας στην ουσία ε, συμβάλλει θα έλεγα σε αυτόν τον αγώνα ανταγωνισμού ανάμεσα στους καπιταλιστές οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν εμπορικά ακόμα και την ίδια της έννοια της ζωή των εμβίων όντων ε, και θέλουν να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου οι εργαζόμενοι να μην ελέγχουν το προϊόν της εργασίας τους και της γνώσης τους. Ξεχνάτε αν θέλετε ότι έχει σχέση και με θέματα εθνικής άμυνας, κάτι το οποίο κάνει τον Αμερικανό νομοθέτη να γελά. Στην ουσία εσείς προχωράτε στην εκμετάλλευση και την πτώση των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, της άκρατης προσπάθειας ιδιωτικοποίησης των πάντων, της υπερβολικής συγκέντρωσης του πλούτου. Οι προτάσεις σας είναι εναντίον της ψηφιακής επανάστασης επίσης. Συνάδελφε, δεν ήθελα να σας διακόψω. Θυμίζω όμως ότι πρέπει να μιλάτε λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουν και οι διερμηνείς μας να σας παρακολουθούν. Ένα λεπτό είναι ένα λεπτό ε, και συγκεκριμένο αριθμό λέξεων μπορείτε να ε, εκφέρετε μέσα σε ένα λεπτό. Ο κύριος Γιόμπρο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Σήμερα συζητούμε μια πολύ σημαντική αλλαγή στο νομικό σύστημα της Ένωσης. Ακούσαμε πολύ αισιόδοξου λόγους κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους πραγματικούς κινδύνους, ε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα καινούργια κράτη-μέλη οι διεθνείς ε, πολυεθνικές ε, προστατεύονται καλύτερα, ιδιαίτερα αν είναι οι Ιαπωνικές, οι Αμερικανικές ή αν προέρχονται από μεγάλα κράτη-μέλη, γιατί το 80% των διπλωμάτων που έχουν ε, απονεμηθεί προέρχονται από αυτές τις εταιρείες αυτού του τύπου. Οπότε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μονοπωλιακή τους θέση ε, με τρόπο κερδοφόρο για αυτές. Θυμίζω ότι πολλέ φορέ οι μεγάλε επιχειρήσει χρησιμοποιούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να μπλοκάρουν την πρόσβαση στην αγορά για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Στην Πολωνία οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη αγορά και σύμφωνα με εκτιμήσεις το κόστος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα αυξηθεί εκθετικά μάλιστα, πράγμα που σημαίνει ότι θα συρρυκνωθεί η οικονομία μας. Αυτές οι απειλές πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Όμπερμαϊρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν το ενιαίο δίπλωμα θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και καινοτόμο δράση της Ευρώπης απέναντι στη ΗΠΑ και την ε, ε, Κίνα θα μπορούσε να φέρει ωφέλη για τις επιχειρήσεις αλλά είμαι επιφυλακτικός για διάφορους λόγους πρώτον σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία ε, ενιαίο ενοποιημένο σύστημα ε, το οποίο θα παραγκώνιζε την τοπική δικαιοδοσία στα κράτη-μέλη και θα ε, ε, επεβάλλεται μόνο το ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, είναι επίσης αμφισβητούμενο το αν θα ήταν αποτελεσματικότερο το σύστημα αυτό. Ε, θα έφτανε στο 25% των εθνικών δικαστηρίων και πολλές φορές οι συζητήσεις θα γίνονταν και κλεισμένων των θυρών. Μου θυμίζει η συζήτηση αυτή της εξελίξης επί άκτα. Επίσης το διαδικαστικό κόστος δεν πρόκειται να το μειώσουμε. Μάλιστα οι ειδικοί υπολογίζουν πλασιασμό του κόστους και των κινδύνων οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θα έχουν την πολυτέλεια να ανταποκριθούν σε όλα αυτά. Οι μεσαίε ε, τάξεις, ε, ε, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται αυτό το σύστημα. Ε, θα πρέπει οι αποφάσεις του... Θα πρέπει να μπορεί κανείς να προσβάλλει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις αποφάσεις του Δικαστηρίου για τα διπλώματα. Και θα πρέπει επίσης να δούμε το θέμα εις ό,τι αφορά τα διπλώματα για ζώα και φυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να είναι εδώ ο κύριος Μπουσουτήλ. Άρα προχωρούμε στην κυρία Μέρκες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συζητητές για μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια την οποία επιτέλεσαν. Μετά από 40 χρόνια επιτέλους οδηγούμεθα μάλλον στο τέλος ενός θέματος ιδιαίτερος περίπλοκου. Το θέμα είναι βέβαια αν τα προτινόμενα μέτρα είναι επαρκή. Το θέμα είναι αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 40 χρόνια δεν μπορέσαμε να λύσουμε το θέμα, τι ακριβώς κάνουμε τώρα. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι καταλήξαμε σε μια πρόταση απόλυτα αποδεκτή από όλους. Δεν έχουμε ένα θησαυρό μπροστά μας. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν, δημιουργούμε ένα σύστημα αρκετά περίπλοκο. Βέβαια το παρόν σύστημα είναι τόσο περίπλοκο που κανένας δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί. Θα έπρεπε όμως να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε αυτό το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευαισθητεχνίας να καλύψει πλήρως τις ανάγκες προώθησης ε, της καινοτομίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλά από αυτά που δεν έγιναν, δεν έγιναν για λόγους δημοσιονομικούς εισαγωγικά και για λόγους προστασίας ε, ε, συμφερόντων. Mr. for one minute, please. Thank you, Chair. Um, I'm very happy that the European patent is, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση μετά από την εκκίνηση εκ νέου της διαδικασίας το 2010. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία να προχωρήσουν σε μια ενιοποιημένη αγορά. Υποτίθεται ότι τώρα έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είπε να απορριφθούν τα αιτήματα και οι ισχυρισμοί της Ιταλίας και της ε, ε, Ισπανίας. Πράγματι έχουμε μειώσει το κόστος της μετάφρασης, το εναρμονισμένο σύστημα αντιμετώπισης των διαφορών ε, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό που κάνουμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καινοτομία και να διευκολύνουμε την ένταξη νέων προϊόντων στην αγορά. Η καινοτομία δεν είναι κάτι το θεωρητικό, είναι κάτι το πρακτικό που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά μας. Ευχαριστώ κύριε Ντεμπάκερ. Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Η, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας υποτίθεται ότι πρέπει να προωθήσει την καινοτομία και να πλουστεύσει την πρόσβαση στην δικαστική προστασία. Αλλά αυτό, ε, αν το πακέτο αυτό το υλοποιήσουμε, οι περισσότερες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να το δεχτούν και χιλιάδες διπλώματα θα ε, καταγράφονται σε άλλες γλώσσες από την γλώσσα της χώρας της επιχείρησης και αν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς στο δικαστήριο σε ξένη γλώσσα, όχι τη μητρική. Θα πληρώνει κανείς περισσότερο για τις μεταφράσεις, θα πληρώνει περισσότερα για τον δικηγόρο και θα δυσκολεύεται η πρόσβαση στην δικαστική προστασία, στην νομική προστασία. Θα φτιάξουμε ένα σύστημα όπου οι ισχυροί θα γίνουν ισχυρότεροι και οι αδύναμοι πιο αδύναμοι ακόμη το σύστημα είναι αντιπαραγωγικό και θα είναι μέσον προστατευτισμού. Οι μικρότερες επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται περισσότερο να έχουν πρόσβαση στην αγορά και αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα περισσότερα διπλώματα ε, ε κατατίθενται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρόβλημα καταλαβαίνετε θα είναι μεγάλο. Κύριε Σφεραίρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να γνωρίζουμε την ανάγκη να προβλεφθεί η διαδικασία για την καταχώρηση του διπλώματος τέχνιας με τρόπο προσιτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για τους εφευρέτες. Όμως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την πρόταση διότι δεν καλύπτει τις ανησυχίες ε, που μας δημιουργεί. Παραδείγματο χάρη, η μεγαλύτερη δημοσίευση, η καλύτερη διανομή των πληροφοριών που είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας ε, προστατεύει τα συμφέροντα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και κάποιων μεγάλων χωρών και δεν εξυπηρετεί ε, το κοινό καλό. Επίσης, ε, ε, χάνουμε την εθνική κυριαρχία με το νέο δικαιοδοτικό σύστημα και είναι προφανής οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Επίσης, ε, υπάρχουν τομείς όπως η κατοχήρωση της ευρεσιτεχνίας για τους ζωντανού οργανισμούς που σε τομείς λοιπόν ευαίσθητους και δεν προβλέπονται οι απαιτούμενες, τα απαιτούμενα ένδικα μέσα για την προβολή ενστάσεων. Συνοψίζονται Τελειώνοντας, ε, αυτή η πρόταση δεν είναι σίγουρα η καλύτερη λύση. Κύριος Πάξας, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υψίσω την προσοχή σας σε κάποια προβλήματα που ενδεχομένως να είναι. Ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, ισχυρίζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την αυτόματη μετάφραση για τις τρεις βασικές ε, γλώσσες, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Ε, όμως αυτό το συζήτημα είναι προβληματικό διότι μπορεί να χρειαστεί τελικά ένας χρόνος για να εξασφαλίσουμε μετάφραση καλής ποιότητας προς περίπλοκες γλώσσες όπως τα λιθουανικά παραδείγματο χάρη. Χώρες όπως η Λιθουανία θα πρέπει να έχουν δικαίωμα για μια μεταβατική περίοδο ώστε οι επιχειρήσεις, ο βιομηχανικός μας κλάδος να μπορέσει να κάνει απαιτούμενες προσαρμογές για ε, το σύστημα αυτό θέμα της ε, μετάφρασης. Επίσης, η δημοσίευση των στοιχείων είναι ε, απαραίτητη και ως εκ τούτου μια επιμελής μετάφραση μπορεί να οδηγήσει σε νομικά προβλήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρία Αντζέλη Κανίμπε, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι δαπανηρό το σύστημά μας, είναι το δεκαπλάσιο σε σχέση με το αμερικανικό και το κινέζικο σύστημα, το είπαν πολύ. Όταν αποφασίσουμε το ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα, αυτό θα είναι ορόσημο στην ιστορία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Ορόσημο, επαναλαμβάνω, στην ιστορία της ολοκλήρωσης της ε, εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό Αρχίζω την παρέμβασή μου με ένα θερμό ευχαριστώ προς όλους τους συναδέλφους, τους εισηγητές πρωτίστως, τους κυρίους Ράπκα, Μπαλτασάρε και Λένε και πολλούς άλλους ε, συναδέλφους που ε, επέδειξαν ενθουσιασμό και που επί δεκαετίες δεν το έβαλαν κάτω παρά τις ήτες των τελευταίων μηνών κυρίως επέμειναν στο ενίο σύστημα με επικοδομητικό πάντα τρόπο και τώρα μπόρεσε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Εγώ είμαι από τη Βαβαρία. Πολλές μικρομεσές επιχειρήσεις εδώ και χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ακούν ότι πρέπει να έρθει μια ενιαία λύση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ε, εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι κινητήρια δύναμη για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θα ψηφίσουμε το μεσημέρι. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απελπισμένα χρειάζονται ένα νέο σύστημα Επίσης, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, εκπαιδεύουν, καταρτίζουν τους νέους. Είναι εκείνοι που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ένωση. Είναι εκείνοι που έχουν το μεγαλύτερο καινοτόμο δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αν αποφασίσουμε αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με λιγότερο κόστος, λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη χρονοβόρο διαδικασία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πραγματικά θα έχουμε κάνει μια σωστή δουλειά. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να υποστηρίξουν το ζήτημα αυτό και στην Επιτροπή Βιομηχανίας κάναμε διαβουλεύσεις ε, για πάρα πολύ καιρό σχετικά με τις προτάσεις ε, της Κομισιόν για το Small Business Act και ένα βασικό θέμα ε, που κολούσαμε είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να έχουν μεταξύ άλλων διότι δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε μέχρι τώρα νομοθεσία νομοθεσία για την ενιαία προστασία του διπλώματος. Βεβαίως ε, ήταν δύσκολη η γένα για το δίπλωμα αυτό. Πολλοί συνάδελφοι ε, μίλησαν για τις εξελίξεις από τη δεκαετία του 70 όπου συζητείται το θέμα, το γλωσσικό καθεστώς ήταν ένα θέμα που είμαι 13 χρόνια στο Κοινοβούλιο και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο από καιρού εις καιρών μας απασχολούσε ε, πολλά χρόνια τώρα. Πάνω από το 90% των διπλωμάτων είναι στα αγγλικά και εγώ ε, ε, δίνω μεγάλη σημασία και αγαπώ τη γλώσσα μου αλλά και τη βαβαρική διάλεκτο πιστεύω παρόλα αυτά ότι το τρίγλωσσο καθεστώς είναι καλό ελπίζω ότι η Ιταλία και η Ισπανία θα περάσουν αυτή την ανοιχτή πόρτα πολύ ωραία το διατύπωσε ο Επίτροπος και θα ε, πραγματικά περιμένουμε να γίνουμε 27 τώρα η έδρα του ενιαίου δικαστηρίου ε, δεν είναι ιδεώδης ε, λύση τώρα με τους τρεις, είναι κλασική περίπτωση αυτή ενός ευρωπαϊκού παραδόξου, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αποφασίσουμε εμείς αυτό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι τα σχόλια στην έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Λένι είναι σωστά, εύστοχα και τελειώνω αναφέροντας κυρίες και κύριοι ότι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού όπως λέμε τόσο ωραία. Αυτό ισχύει και για το ενιαίο δίπλωμα τεχνίας. Ελπίζω ότι με μεγάλη πλειοψηφία θα ε, εγκρίνουμε και θα θεσμοθετήσουμε κάτι που περιμέναμε πολλά χρόνια. Ε, τις ε, προτάσεις εγώ θα τις υπερψηφίσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπένοβα, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το ενιαίο σύστημα θα υπάρχει παράλληλα με τα εθνικά συστήματα, ε, αυτό το περιμέναμε χρόνια. Τώρα με την έγκριση των προτάσεων όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προστατεύουν και να κατοχυρώνουν τις εφευρέσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το υψηλό κόστος είναι το, ο βασικός λόγος για τους οποίους οι ιδιοκτήτες των διπλωμάτων δεν επίπεδίωκαν ε, ευρωπαϊκή προστασία. Το κόστος ανέρχεται σε 22 με 26 ευρώ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διπλωμάτων ε, θα ε, στοιχίζει 680 ευρώ μόνο και θα προσφέρει καλύτερα, καλύτερες προϋποθέσεις. Θα είναι απλούστερο το ευρωπαϊκό σύστημα και οι χρήστες τις διαδικαστικές τους δαπάνες θα μπορέσουν να τις μειώσουν κατά 80% περίπου, μέχρι και 80%. Έτσι η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά θα διασφαλίζεται και θα μπορούμε τις επενδύσεις μας στην έρευνα και την ανάπτυξη του 3% του ΑΕΠ να τις ε, υλοποιούμε όπως προβλέπεται στη στρατηγική 2020. Επίσης θα υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου στο ζήτημα αυτό. Προσθέτω ότι το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα θέματα. παρακαλώ για λεπτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή ή τους εισηγητές για την εξαιρετική τους δουλειά. Θα ήθελα όμως κυρίως να συγχαρώ τον κύριο Μπαρνιέ. Μετά από μια συζήτηση που κράτησε 40 χρόνια, καταφέρατε να μας οδηγήσετε στο τέλος του δρόμου. Σας ευχαριστώ για αυτό και εξ ονόματος της περιοχής ε, του Ολλανδικού Μπράμπαντ που παρουσιάζει τέσσερις αιτήσει την ημέρα για χορήγηση διπλωμάτων ευαισθητεχνίας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εγώ είχα καταθέσει επαγγελματικά παλαιότερα κάποιες αιτήσει για χορήγηση τέτοιων διπλωμάτων αλλά σε επίπεδο Μπενελούξ όπως ήταν κάτι τέτοιο εφικτό γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Είναι σημαντικό αυτό που έγινε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για την δυνατότητα υιοθέτηση αυτής της προσπάθειας. Λυπάμαι που δύο χώρες δεν συμμετέχουν στο σύστημα. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα εργαστήκαμε κάτω από ένα σύστημα το οποίο δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό και τώρα είναι κρίμα που δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Μάντερς. Κύριος Τοσενόφσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας έχει φτάσει πλέον στην τελική του φάση. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια επιπλέον όθηση στην τόσο επιθυμητή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το τσεχικό επιμελητήριο, εμπορικό επιμελητήριο είναι ικανοποιημένο από τις προτάσεις αυτές. Αυτό ε, που πρέπει να γίνει τώρα είναι να υπάρξει μια σωστή εφαρμογή αυτών των μέτρων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα λειτουργικό σύστημα, ένα σύστημα διοικητικά απλό, ένα σύστημα διεθνώς αποδεκτό. Γνωρίζουμε τώρα ότι πολλές φορές βέβαια οι καλές προθέσεις λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας δεν ικανοποιούν. Το παρακαλώ. Κύριε Σαγκουράκη. Στόχος του ενωσιακού συστήματος ευρεσιτεχνίας είναι η παραπέρα ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων στην ενιαία καπιταλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια στις παγκόσμιες αγορές με φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου των προϊόντων πνευματικής δημιουργίας. Αυτό θα εντείνει τη συγκέντρωση των ευρεσιτεχνιών στα χέρια οικονομικά ισχυρών ομίλων και θα ενισχύσει την μονοπόληση της γνώση όπω ακριβώ επιτάσσουν οι πιο ισχυρέ πολυεθνικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση των εργαζομένων σε προϊόντα και υπηρεσίε σε κρίσιμου τομεί όπω την υγεία τα φάρμακα ενέργεια τρόφιμα κλπ που σε ακόμα μεγαλύτερη έκταση θα αποτελούν αντικείμενο καπιταλιστική κερδοσκοπία. θεσμοθετείται με το σύστημα αυτό ένα νέο δικαστικό σύστημα για τις ευρεσιτεχνίες που θα κρίνει με βάση ένα συνοθήλευμα ακόμα πιο αντιδραστικών νομικών διατάξεων που υπερισχύουν του εθνικού δικαίου. παρακάμπτονται έτσι μια σειρά περιορισμοί στην έκταση των ευρεσιτεχνιών που προβλέπονται σήμερα από το εθνικό δίκαιο. έτσι όμω δημόσια κοινωνικά αγαθά και επιστημονικά επιτεύγματα θα εμπορευματοποιούνται όλο περισσότερο και δεν θα είναι προσβάσιμα. ευχαριστώ. Εγώ, ο Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα σίγουρα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για να χαμηλώσει το κόστος το οποίο είναι απαραίτητο για τις μεταφράσεις και τις καταγραφές ε, των διπλωμάτων αυτών. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις, θα γλιτώσουν κάποιες χιλιάδες ε, ευρώ. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης όπως ε, η τωρινή, αυτό είναι σημαντικό έπρεπε ίσως να επιλεγεί μία γλώσσα η οποία για διάφορους λόγους δεν μπορεί παρά να είναι τα αγγλικά. Αυτός, αυτή η τριγλωσία είναι προκλητική. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα γαλλικά και τα γερμανικά θα πρέπει να ευνοούνται σε σχέση με τις υπόλοιπες. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόσφατα έχει απορρίψει για τους διαγωνισμούς έψω αυτή τη φόρμουλα σε τρεις γλώσσες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα. Καλό είναι να εξοικονομούμε χρήματα, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χάνουμε την ώρα μας και τα λεφτά σε μεταφράσεις γαλλικά και γερμανικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως υπενθύμησαν και οι συνάδελφοί μου, 40 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια περιμένει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεστεχνίας η Ευρώπη. Τώρα το ζούμε, ζούμε μια ιστορική στιγμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μπάρνιε είναι απαραίτητο αυτό το νέο εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας ε, των επενδύσεων ε, στην έρευνα και την καινοτομία από πλευρά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται την καινοτομία, χρειάζεται τι εφευρέσει ε, και το δημιουργικό κλίμα, διότι δεν είναι ικανοποιητικέ οι αποδόσει μα. 60.000 διπλώματα κατατίθενται στην Ευρώπη, έναντι 172.000 στην Κίνα και 224.000 στι ΗΠΑ. Ε, χάνουμε τώρα το τυπάχι και πρέπει να αντιδράσουμε. Το πακέτο όπου θα εγκρίθει αμφισβητείται από διάφορους βουλευτές και πανεπιστημιακούς καθηγητές. Ισχυρίζονται ότι το νομοθετικό πλαίσιο που τώρα θεσπίζουμε δεν είναι τέλειο. Ε, δέχομαι και ασθενίζομαι κάποιες από τις επικρίσεις τους, όμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία λόγω αυτών των ακαδημαϊκών συζητήσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι η επίπτωση ε, του νομοθετήματο αυτού για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η προστασία, η νέα προστασία μέσω του διπλώματο ε, θα μειώσει έξι φορές ε, το κόστος από 30.000 Από 30.000 θα περάσουμε στις 5.000 ε, για το κόστος ε, του διπλώματος. Θα ενισχύσουμε έτσι την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι να θεσπιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο ενιαίας προστασίας ε, που θα εδράζεται στη μέχρι τούδε πρακτική του Ευρωπαϊκού Γραφείου ε, που έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αισίως και επίσης επί της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της απόφασης 8 Μαρτίου 2012 σχετικά με τα διπλώματα. Επίσης εν τέλει πρέπει να υπερβούμε τη δυσκολία του άρθρου 118 της συνθήκης της Λισαβόνας που απαιτεί την ομοφωνία στο Συμβούλιο για τα γλωσσικά ε, κάθε εστότα των νέων τίτλων εκατοχήρωσης ε, διανοητικών δικαιωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τις πολιτικές και νομικές δυσκολίες ε, στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε, πιστεύω ότι αυτό είναι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα της διαδικασίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόθερμα τους κυρίους Ραπκάη, Μπαλτασάρη και Λένα για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, την υπομονή που έδειξαν και την ευούληση να καταλήξουν σε συμβαστική λύση. Ας δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ας παρατηρήσουμε την λειτουργία του, διαπιστώσουμε ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του και ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει πάντοτε τη δυνατότητα να επιφέρει βελτιώσεις ή τροποποιήσεις σε αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο μελλοντικά. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ελπίδα η Ισπανία και η Ιταλία να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να συμμετάσχουν πλήρως στο ε, σύστημα ενιαίας προστασίας μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε καταπληκτική ευκαιρία για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και ενάπτυξης. Θα Σας ευχαριστούμε κύριος Λούντβιξον τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι θετικό που τελικά ε, θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ευρωπαϊκό Σύστημα Κατοχήριωση ε, μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ε, καλές οι επιδόσεις, βελτιώνεται το σύστημα και απλουστεύεται η διαδικασία και επίσης γίνονται φινότερα τα διπλώματα. Ισχύουν καλύτεροι όροι για τις καινοτόμες ευρωπαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται και προστατεύονται ε, σε σχέση με τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτό είναι σημαντικό, τόσο ώστε η Ευρωπή να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να τονώσει ε, την ανάπτυξή της Και εδώ και καιρό δεν είχαμε δει τέτοια ευκαιρία, αναπτυξιακή ευκαιρία όπως τα διπλώματα έβρεση τεχνίας. Ε, μέσα στο πακέτο αυτό υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν ε, κάποιες θεμητές ανησυχίες. Δεν είναι ιδανική λύση, αλλά είναι καλή συμβαστική λύση ε, δεδομένων των δυσκολιών που είχαμε. Εξισορροπείται έτσι το νέο σύστημα κατοχύρωσης ε, μέσω ενός νέου νομικού πλαισίου και άρα θα μπορέσουν να προσυπογράψω. Επιτέλους ε, περνάμε από τα λόγια στις πράξεις ε, για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Today is going to be... Σήμερα θα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ευρώπη, τους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μετά από 40 χρόνια διαπραγματεύσεων Έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ισχυρό για τις περισσότερες χώρες για την προώθηση της ενιαίας αγοράς. Όμως η Ισπανία αρνείται να συνδεθεί με αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο. Μου δημιουργεί μια δυστημία γιατί για λόγους εθνικιστικούς χαμηλού επίπεδου η Ισπανία αρνείται να συμμετέχει χιλιάδες ανταγωνιστικές ισπανικές επιχειρήσεις ε, θα φυγούν από αυτήν την εξαίρεση. Εγώ είμαι Καταλανός, προέρχομαι από την Καταλωνία. Το 30% των ισπανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι από την Καταλωνία. Η στάση της Ισπανίας είναι απαράδεκτη. Εγώ θα στηρίξω το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, βελτιώνοντας την ενιαία αγορά, βελτιώνουμε τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Η ισπανική κυβέρνηση δίνει κίνητρα και κυρίως δίνει επιχειρήματα για να ζητήσουμε να δημιουργηθεί ένα νέο ανεξάρτητο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Τεμόζα. Ιμπαλσέλς. Έχετε μία μπλε κάρτα. Την δέχεστε. Από τον κύριο Λόπες Ιστούρης. Δέχεστε μία μπλε κάρτα. Μιλώντας για εθνικισμούς, Πολλές φορές μιλάμε με αρνητικό τρόπο και θα πρέπει να εξηγήσουμε στους καταναλούς, κα, ε, καταλανούς φίλους ότι προβλέπεται ένα γλωσσικό σύστημα το οποίο δεν είναι φυσικά, δεν περιλαμβάνει τη γλώσσα τους, δεν περιλαμβάνει ούτε την ισπανική γλώσσα και γι' αυτό όταν μιλάμε για εθνικιστικές χρήσεις των γλωσσών στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα πρέπει να μιλάμε για την Ισπανία, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ανταπαντά ο κύριος Μπασέλς στον Λόπες Ιστούρης. Τα αγγλικά είναι και αυτή δική μας γλώσσα. Στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης τα υπάρχουν μαθήματα και στα καταλανικά και στα αγγλικά. Αυτό δεν δημιουργεί στις καταλανικές επιχειρήσεις που εξάγουν περισσότερο στις ευρωπαϊκές χώρες παρά στην υπόλοιπη Ισπανία. Ε, το να χρησιμοποιούμε τα αγγλικά είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει κατά πολύ τη διαχείριση των συστημάτων και τη ροή των συναλλαγών και της καινοτομίες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, το να μην υποστηρίζει κανείς ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι σαν να πηγαίνει ενάντια στα συμφέροντα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μασίπη Δάλγο θέλει και αυτός να σας θέσει ένα ερώτημα με μπλε κάρτα. Δέχεστε το ερώτημα. Κύριε Μπασέλς. Έχετε και άλλη μία ερώτηση. Signor Ντάρκο. Ακούμε εδώ ότι ο εθνικισμός λειτουργεί εις βάρος των επιχειρήσεων. Οπότε κύριε Τρεμόσα εσείς γιατί δεν απαρνείστε τον εθνικισμό ο οποίος επηρεάζει τόσο άσχημα τις καταλανικές επιχειρήσεις. Bien, Απαντώ στον φίλο μου τον κύριο Μασίπ λέγοντας ότι εγώ είμαι καταλανός αισθάνομαι Ευρωπαίος Καταλανός. Και να πω ότι η καταλανική οικονομία, άλλωστε μετά από τις τελευταίες εκλογές θυμίζω ότι τα δύο τρίτα των εκλογέων ψήφισαν για κόμματα τα οποία θέλουν να κάνουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, πιστεύουμε ότι στην ουσία Υπάρχουν χιλιάδες επαγγελματιών οι οποίοι εξάγουν τα προϊόντα τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και από το σύνολο της Ισπανίας. Ε, μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν προς όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα να σεβόμαστε σαν λαό την ταυτότητά μας και τις ρίζες μας. Για ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ. Ο Winston Churchill είπε κάποτε ότι όποτε είχα δίκιο ήμουν στη μειοψηφία. Και εγώ ήμουν στη μειοψηφία όταν μιλούσαμε για τη μεταρρύθμιση ε, του... Και σήμερα ε, είμαι στη μειοψηφία κρίνοντας ε, αυτά που ακούσαμε γιατί είμαι κατά του συστήματος και είμαι κατά γιατί στη χώρα μου την Πολωνία αυτό το εγχείρημα απερίφθη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από επιστήμονες, από την κοινωνία γενικότερα γιατί όλοι βλέπουν ότι το κόστος θα αυξηθεί για να πάρει κανείς το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ιδιαίτερα θα αυξηθεί το κόστος για τις μικρομεσαίες ε, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη χώρα μου βλέπουν ότι έτσι προστατεύουμε τα συμφέροντα των μεγάλων και βλάπτουμε τα συμφέροντα των μικρών οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα και νομίζω ότι ε, για τις βιολογικές διαδικασίες τα διπλώματα θα είναι ε, εναντίον της γεωργίας η οποία θα αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη τομέας της οικονομίας. Εγώ είμαι κατά και θα το καταψηφίσω. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην αίθουσα αυτή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα μιλάμε όλοι για την βελτίωση και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, την ανάγκη για οικονομική μεγέθυνση ανάπτυξη, γιατί χωρίς οικονομική ανάπτυξη η Ευρώπη θα χάσει χρήματα και δεν θα έχει πια κεφάλαια για την διατήρηση των δαπανηρών κοινωνικών συστημάτων. Το θέμα είναι πώς θα την κατακτήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις μας ε, θα ε, εφαρμόσουν δημοσιονομική πειθαρχία για να τα επιτύχουν όλα αυτά. Υπάρχουν επίσης και μεγάλες ε, δυνατότητες μέσα από την νομοθεσία διότι έτσι θα ε, ενισχυθεί το εργατικό δυναμικό εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη και σε έφθετο χρόνο πρέπει να έχουμε ετοιμάσει, καταρτήσει το ανθρώπινο δυναμικό μας ούτως ώστε να ε, αυξηθούν τα ε, έσοδα. Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι για το μέλλον αυτών των ανθρώπων ε, πρέπει να διασφαλιστούν και τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν προβλήματα με το σύστημα επίλυση διαφορών, με τα γλωσσικά καθεστώτα κλπ. Λύσει υπάρχουν και αυτέ μα απασχολούν σήμερα. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, μετά από περίπου 40 χρόνια διαπραγματεύσεων, επιτέλου φτάσαμε σε ένα στάδιο στην Ευρώπη όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο σύστημα προστασία διπλωμάτων. Δεν είναι τέλειο το σύστημα. Δύο χώρε, Ισπανία και Ιταλία, ακόμη δεν επιθυμούν να ε, ενταχθούν. Στα 25 κράτη-μέλη όμως, αν μια νέα εταιρεία, ένας νέος εφευρέτης ή παλαιός εφευρέτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την απλουστευμένη διαδικασία για ε, ενιαίο δίπλωμα το οποίο εξασφαλίζει προστασία σε 25 κράτη-μέλη, αυτό είναι πολύ καλό. Στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία ε, αυτό το σύστημα είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος. Τώρα είναι η ευκαιρία να ε, αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν είναι η τέλεια λύση, το επαναλαμβάνω, αλλά είναι μια καλή λύση που θα δώσει, θα αποτελέσει μια βάση, ένα θεμέλιο για το μέλλον της ανάπτυξής μας. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εφευρέτες μας που θα βοηθήσουν με τη σειρά του την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, πράγματι έχουμε να κάνουμε... Έχουμε να κάνουμε με μια πλήρη πολυδιάσπαση της αγοράς. Θέλουμε αποτελεσματική χρήση ε, των διπλωμάτων για τις, Ευρωπα... για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε έτσι να εδρεώσουμε τις εφευρέσεις στην Ευρώπη. Ένα ενιαίο δίπλωμα μπορεί να βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη ή κάποια κράτη-μέλη. Το ενιαίο σύστημα θα μειώσει και το κόστος για τους ετούντες κατά περίπου 70%. Τα τέλη ανανέωσης ε, θα ε, προσδιοριστούν, θα καθοριστούν λαμβάνοντας ε, υπόψη και την ιδιαιτερότητα των μικρομεσαίων. Και το η γλωσσική ρύθμιση είναι σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη και επίσης και το κόστος για τις μεταφράσεις. Οι μηχανικές μεταφράσεις, οι αυτόματες μεταφράσεις ακόμα βέβαια δεν έχουν την νομική ακρίβεια που χρειάζεται. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένα τμήμα για την ανατολική Ευρώπη γι' αυτό, για το ενιαίο αυτό σύστημα. Κυρία Ρης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Είναι ιστορική σημασία η εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μετά από 30 χρόνια, 30 χρόνια συγγνώμη, υπερβαίνουμε τις ε, άγονες αντιπαραθέσεις και θεσπίζουμε ένα νέο σύστημα προστασίας των εφευρέσεων, εξυπηρετώντας το έργο της μείωσης του κόστους. 30.000 ήταν το κόστος ε, σε 10 χρόνια, τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος, 10 ε, φορές περισσότερο από τη ΣΥΠΑ την Ιαπωνία. Δεν ξέρω κύριο Στασκόφσκι που τα βρήκε αυτά τα στοιχεία. Το πρώτο δίπλωμα που θα μπορέσει να κατατεθεί το 2014 θα κοστίζει 5.000 για τους εφευρέτες και έτσι θα μπορέσουν να αποφύγουν αυτό τον ανώμαλο δρόμο που διέσχιζαν για κατοχυρώσουν τις εφευρέσεις τους ε, ε, και να ε, ανακάμψει το ηθικό των εφευρετών και των επιχειρήσεων χρειάζονται και άλλες προσπάθειες αλλά το δίπλωμα είναι θεμελιώδης σημασία όμως δεν επαρκεί. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται καλύτερη βιομηχανική προστασία όμως ταυτόχρονα χρειάζονται και κεφάλαια, διευκολυμμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον περιβάλλον, ε, ούτω ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε. Μασίπ Χιντάλκο Αντώνιο. Presidenta, bien lo siento, pero no es patente. Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένα ευρωπαϊκό θα έλεγα σύστημα ευρεσιτεχνία. Γίνεται διάκριση εις βάρος των Ισπανών υπέρ της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσας. Δημιουργούνται επιπλέον κόστη και στην ουσία ε, περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Τα άρθρα 8, ε, 6 και 7 δεν είναι διόλου ικανοποιητικά. Δημιουργείται ένα σύστημα νομικής δικαιοδοσίας το οποίο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Πρέπει να είμαστε λιγότερο ε, πανηγυρικοί στον τρόπο που παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα αυτό και να μην μένουμε στην παρουσία την οποία έκανε ο Γενικός Εισαγγελέας στο δικαστήριο. Η κυρία Καστέξ δεν είναι παρούσα. Ε, στον κύριο Ρέπο. Κυρία Πρόεδρε, Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τους συναδέλφους. Θέλω και εγώ να τονίσω τη σημασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο αριθμός των διπλωμάτων και η προστασία των άλλων δικαιωμάτων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ένας λόγος είναι ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται όλο και περισσότερο στην καινοτομία. Τα τελευταία χρόνια περίπου το 80% όλων των νέων θέσεων εργασίας ε, δημιουργήθηκαν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πολύ λίγε μικρές, μικρομεσαίες ζητούνται ε, δίπλωμα για τα προϊόντα τους όμως και ένας λόγος πάλι είναι ότι στην χώρα τους λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου ε, τα άειλα δικαιώματα δεν έχουν μεγάλη σημασία. Οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύσκολα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ε, ιδιαίτερα επειδή θα είναι πιο δαπανηρό ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα που θα ετηθεί ε, σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον θέλουμε να λειτουργεί καλά η εσωτερική αγορά. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνία είναι πολύ σημαντικά και για τη στρατηγική 2020, Ευρώπη 2020, γιατί τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και έμεσα δημιουργούν απασχόληση. Κόβατ επίση δεν είναι στην αίθουσα, οπότε περνάμε στην διαδικασία Catch και θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλη. Μετά από 60 χρόνια προσπαθειών πήραμε τον Νομπέλ Ειρήνης, καταπληκτικό επίτευγμα. Και σήμερα μετά από πάνω από 30 χρόνια ε, έχουμε αυτό που θα αποκαλούσαμε σε εισαγωγικά ενιαίο σύστημα προστασίας. Ε, κάποιοι δεν επιχαίρουν ε, ακούσαμε ότι αυτά που μας είπε ο Επίτροπος Μπαρνιέ είναι δυναμική αυτή η συμβαστική λύση. Εάν τονώνει την ανταγωνιστικότητα, προφανέστατα είναι καλό το σύστημα. Αν αυξήσει τον αριθμό των διπλωμάτων, αυτό θα είναι απόδειξη της επιτυχίας του συστήματος. Όπως είπε η κυρία Γκάλο, 60.000 περίπου διπλώματα κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σημειωθεί αύξηση, τότε θα σημειωθεί και πρόοδος. Ε, είναι προφανές ότι θα θέλαμε να προσχωρήσουν και η Ιταλία και η Ισπανία και θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο Μπαρνιέ να μεριμνήσει ούτω ώστε να γίνει αυτό και πώ σκοπεύει να το κάνει. Υπάρχουν, γίνονται συγκεκριμένε προσπάθειε. Ο κύριο Τσφέρ. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Ε, με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές ε, Ραπκάη, Λένε και Μπαλτασάρη Συγχαρητήρια προς τον Επίτροπο Μπαρνιέ επίσης. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία ε, διότι χάνει το δυναμικό της ρυθμός της ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπορικές συναλλαγές η Ευρώπη. Δεν είμαστε επαρκώς καινοτόμοι όπως το παρελθόν. Αυτό θα επηρεάσει την πρόοδο των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο σύστημα θα επιτρέψει στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν βήματα προς τα μπροστά, θα μειωθεί το κόστος και θα είναι ασφαλέστερα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επίτροποι, υποστηρίζω το έργο σας και όπως και εσείς ε, θλίβομαι διότι διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων τα σλοβενικά, η γλώσσα μου δεν θα έχουν ισότιμη θέση. Εάν όμω, το, το μη χειρον βέλτιστον όπως λέμε και φυσικά θα επιλέξω την ευρωπαϊκή οδό παρά, παρά το ότι υπάρχει αυτό το μειονέκτημα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα έτσι για την ε, επίλυση των διαφορών. Και ένα τέτοιο δικαστήριο είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά την εφαρμογή του λογισμικού. Και εκεί η απονομή των διπλωμάτων διαφέρει, είναι που διαφέρει μεταξύ των χωρών. Νομίζω, σε σχέση με τις δομές που θα ασχολούνται, ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την προστασία νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα σε εφαρμογές λογισμικού, για να έχουμε καλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να αποφύγουμε τις ε, ενστάσεις και τις αμφισβητήσεις. Επίσης είναι σημαντικό για το μέλλον να προσέξουμε την ποιότητα των μεταφράσεων και να έχουμε ειδικού για τις μεταφράσεις αυτές. Προγράμματα αυτόματης μετάφρασης δεν αρκούν για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ποιότητα σε τέτοια ειδική ορολογία. Ευχαριστώ. Επίτροπος Μπαρνιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μπορώ να είμαι σύντομος, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εξέφρασαν τις απόψεις τους με ειλικρίνεια. Ενδεχομένως επιγραμματικά θα ε, ήταν καλό να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η κυρία Λίχτεμπεργκε αναφέρθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρέμβασή της, υποδεικνύοντας ότι βγαίνει από το παιχνίδι το δικαστήριο. Ειλικρινά δεν ισχύει αυτό. Το δικαστήριο ε, θα αποφαίνεται ε, για τα διπλώματα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο άρθρο. Το ίδιο ισχύει για τις μεταφράσεις. Επίτροπε διακόπτη πρόοδος. Έχουμε ένα πρόβλημα με την γερμανική μετάφραση. Ένα λεπτάκι. Θα ξαναρχίσω από την αρχή. Ε, κυρία Λίχτεμπεργκερ. Για να μην υπάρξει παρανόηση, σας επιβεβαιώνω ότι σε τελευταίο δικαιοδοτικό βαθμό το δικαστήριο θα ερμηνεύσει ε, όλο το διατακτικό της απόφασης ε, για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το ίδιο θα ισχύει και για τις μεταφράσεις. Οπότε το νέο σύστημα νέας προστασίας προστατεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως και τα Εθνικά Δικαστήρια, έτσι και το Δικαστήριο ε, της Ένωσης ε, θα επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων ερμηνείας ε, των δύο κανονισμών. Δεν τελειώνει εδώ η διαδικασία. Η κυρία Ρίς μας είπε ότι είναι μία αναγκαία αλλά όχι επαρκής πρόοδος. Θα συμφωνήσω. Θεσπίζουμε το πλαίσιο και τώρα θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω τις λειτουργικές διατάξεις με τρόπο ώστε την Άνοιξη του 2014 να είναι πλέον λειτουργικό ε, το σύστημα και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε αυτό το ενιαίο δίπλωμα σε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση με το που θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα. Ε, κυρία Βίξτρομ, ε, Καρύμ, Γκαλό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους Έχω τη θέση του Επιτρόπου, γνωρίζετε και εδώ και χρόνια συνεργάζομαι με το επιτελείο για αυτό το θέμα. Όλες οι διαδοχικές προεδρίες από τη Γαλλική, την Βελική μέχρι και την Κυπριακή, την οποία ευχαρίστησα στην ανακτήρια παρέμβασή μου, ε, να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές ε, του Κοινοβουλίου, ε, λένε Μπαλταζάρη Ράπκαη, ε, ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα του γλωσσικού καθεστώτος, το οποίο ε, είναι δύσκολο. αλλά εξ αρχής σεβόσασταν τον απότερο στόχο μας που είναι να είναι κοινοφελές το, το, το νέο σύστημα. Ο κύριος Ιντάλγο εξέφρασε επίσης θεμητές απόψεις. Μένει ορθά ανοιχτή η πόρτα για την Ιταλία και την Ισπανία. Ο κύριος Κέλλη με ρώτησε πότε. Πότε θα προσχωρήσει η Ιταλία και η Ισπανία στο σύστημα. Ε, είναι δική τους επιλογή, κυρίαρχα κράτη είναι και ε, αυτή είναι η φιλοσοφία της ενισχυμένης συνεργασίας, ότι παραμένει ανοιχτή η πόρτα για όλους τους ε, υπολείπους. Ε, βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νομολογία του δικαστηρίου που περιμένουμε με σεβασμό αλλά και πεποίθηση ότι ε, θα υποστηρίξουν τις αποφάσεις μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την προσήλωση και την αφοσίωσή σας. Ε, ε, απευθύνω σε ευχαριστίες μου στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο αλλά και στην Επιτροπή. Συνιστά ουσιαστική πρόοδο για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη το βήμα που κάνουμε σήμερα και είναι κυρίως ευνοϊκό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μια τελευταία παρατήρηση δεν κατανοώ αυτό που είπαν ο κύριος Σιμάσκι ή ο κύριος Ενά. Ε, βλέπετε στις δύο ακραίες πτέρυγες του ημικυκλίου. Ε, δεν θα ενισχύσουμε τους κρατεότερους και θα αποδυναμώσουμε τους ασθενέστερους. Όχι, δεν είναι ευσταθεί αυτό. Ε, δημιουργείται μια δυναμική ε, μέσω του νέου συστήματος θα είχα και εγώ προκρίνει με διαφορετική μέθοδο, σας το είπα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι προστατευμένες. Ο κύριος Μάντερ είπε πριν ε, πως ότι όταν ήμουν εγώ εφευρέτης δεν προστατεύτηκα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έπρεπε να εκταμιεύσω 25-30 χιλιάδες, μα θα μειωθεί το κόστος, θα απλουστεύσουμε τα διαβήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θετικό για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε. διότι μην ξεχνάτε ότι από τα 22 εκατομμύρια επιχειρήσει, τα 21 εκατομμύρια είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όντως θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Ευχαριστώ. And on behalf uh, of the... Και τώρα από πλευρά της Κυπριακής ε, Προεδρίας και του Συμβουλίου ο κύριος Λουκά. αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός πως τόσοι πολλοί εδώ αυτό το πρωινό μοιράζονται την άποψη του Συμβουλίου ότι είναι καιρός να ολοκληρωθεί το θέμα του πακέτου για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ένα, ένα ενιαίο σύστημα διπλω, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συνέχισης των προσπαθειών μας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και θα βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Το θέμα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και χρειάστηκε αρκετός χρόνος και ενέργεια για να ολοκληρωθεί. Τόσο οι προηγούμενες Προεδρίες όσο και η Κυπριακή Προεδρία κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι η δουλειά αυτή αποδίδει καρπούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωκοινοβούλιο για την κατανόησή του και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μαζί σε αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ. Υπουργέ, και τώρα θα περάσουμε στους εισηγητές και πρώτα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λίνε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους όσους συμμετέσχουν σε αυτή την επικοδομητική συζήτηση ε, και, και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις σωστές διευκρινήσεις. Είναι τεράστια η πρόοδος για τις μικρομεσαίες να σας το πω με ένα παράδειγμα. Σήμερα, χωρίς αυτό το πακέτο ε, και ε, χωρίς ε, το νέο δίπλωμα και το δικαστικό σύστημα, αν ένας μικρομεσαίος ζητήσει δίπλωμα, ακριβή υπόθεση αυτή, και περιορισμένοι μόνο μπορούν να κάνουν την αίτηση, και αν θέλει να επιβάλλει το δίπλωμα απέναντι σε κάποιον που θα το παραδιάσει ε, θα πρέπει να προσφύγει σε 25 κράτη-μέλη. Αυτό βεβαίως ε, θα τον φέρει στα όρια της επιβίωσης του τον μικρομεσαίο. Πρακτικά, συχνά, στην πράξη, ε, συχνά ο μικρομεσαίος θα αναγκαστεί να κλείσει μια συμφωνία ε, ούτως ώστε να μην ζημιώσει πολύ. Εάν ένας μεγάλος επιχειρηματίας ε, κάνει παραβίαση ε, μπορεί να επιβιώσει σε 25 ε, ξεχωριστές χώρες μέλη ε, σε βάρος του μικρού. Έτσι λοιπόν τώρα μπορεί ο μικρός επιχειρηματίας με ένα σύστημα, ένα ενιαίο σύστημα να το χρησιμοποιήσει και αυτό να ισχύει και στα 25 κράτη-μέλη. Για πρώτη φορά λοιπόν θα έχουν τα ίδια όπλα οι μεγάλοι και οι μικροί. Και αυτό για μένα είναι πολύ καθοριστικό για να κρίνω ότι πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα μπροστά αυτό που αποφασίζουμε σήμερα για τους μικρομεσαίους. Και πολλά από αυτά που ακούσαμε προς διαφορετική κατεύθυνση είναι νοησίες για να το πούμε καθαρά. Κανεί δεν υφίσταται διακρίσει γιατί η Ισπανία και η Ιταλία εξακολουθούν να συμμετέχουν στη συμφωνία ε, όλες οι, όλα τα διπλώματα που ισχύουν δηλαδή στην Ισπανία και την Ιταλία θα μπορούν να μεταφράζονται στι απαραίτητε γλώσσε. Το νέο σύστημα δεν αντικαθιστά το παλιό. επίση αντίθετα ε, δημιουργεί μια νέα ακόμα δυνατότητα. Ε, σε σχέση με τα εθνικά διπλώματα, το ευρωπαϊκό δίπλωμα, υπάρχει εδώ μια πρόσθετη δυνατότητα που διευρύνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά είναι από τα σημαντικότερα νομοθετήματά μας κατά τη διάρκεια της θητείας μας και αν αποφασιστεί αυτό θα κάνει η Ευρώπη ένα μεγάλο βήμα μπροστά συνολικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Λίνε και θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Πάλτα Σάρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν το λόγο. Να ήθελα να αναφερθώ σε μια φράση στην οποία αναφέρεται ο κύριος Λένε συχνά «Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού». Νομίζω ότι αυτό ήταν, θα έλεγα, το χαρακτηριστικό όλων των παρεμβάσεων, ακόμα και αυτές οι οποίες άσκησαν κριτική. Έχουμε ένα θετικό, θετικό επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι θα έπρεπε να είχαμε ή θα μπορούσαμε να είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως αυτό έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη ουσιαστική μείωση του κόστους, σε βάθος μείωση του κόστους και στην πρώτη φάση και στη διαδοχική φάση, τη νομική φάση αν θέλετε. Έχουμε μια ρύθμιση που θα ισχύει για 25 χώρες, ελπίζω σύντομα σε 26 και μετά σε 27. Έχουμε ένα τρίγλωσσο σύστημα ε, κοιτάξτε κύριε Μοργάντη και εγώ είμαι πεπισμένος ότι τα Ιταλικά είναι η πιο μουσική και πιο όμορφη γλώσσα στον κόσμο, η πιο αρμονική γλώσσα στον κόσμο. Αλλά αν το 45% των επιχειρήσεων θέλουν να καταγράφονται στα αγγλικά και οι δικοί μας επιχειρηματίες, οι Ιταλοί καταθέτουν τις αιτήσει τους ε, κατά 50% ε, στα αγγλικά, και στο 90% των νομικών διαδικασιών επιλέγουν τα αγγλικά, τότε πραγματικά δεν θα πρέπει να δίνουμε μάχης επί της αρχής, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τις Ιταλικές επιχειρήσεις. Έχω εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα αυτού του συμβιβαστικού πακέτου και θα πρέπει να περάσουμε σε ε, έλεγχο της ενιαίας πλέον εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων με μια μεταβατική περίοδο που θα, εφαρμόσει, που θα εφαρμοστεί έτσι ώστε να δώσει χρόνο στις επιχειρήσεις να συνδεθούν καλύτερα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, να γνωρίσουν σωστότερα το σύστημα των μεταφράσεων, να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα το ευρωπαϊκό πλέον, είναι κάτι το θετικό και ελπίζω ότι και η χώρα μου θα ακολουθήσει μία γραμμή η οποία ε, θα έλεγα είναι διαφορετική από αυτήν που ακολουθεί σήμερα γιατί δεν έχει νόημα να δίνουμε μάχες ε, επί της αρχής όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Ράπκαη. Κυρία Πρόεδρε, έχει δίκιο ο συνάδελφος Μπαλταζάρε και εγώ θεωρώ ότι τα Ιταλικά είναι η ωραιότερη γλώσσα και το λέω αυτός Γερμανός. Αλλά εδώ δεν είναι καλυστία, δεν αποδίδουμε βραβεία ομορφιάς της γλώσσας, εδώ πρόκειται για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τις μικρομεσαίες επιτέλους να εξυπηρετηθούν. Εγώ είμαι πάνω από 18 χρόνια στο Κοινοβούλιο και σπάνια παρευρέθην σε συζήτηση όπου οι αντίπαλοι ενός επιχειρήματος περιέπεσαν σε τόσες αντιφάσεις και μάλιστα πολλοί ε, ε, έπεσαν και σε εσωτερικές αντιφάσεις. Ο συνάδελφος Λόπες δύο φορές μέσα σε μία φράση κατάφερε να ε, παρουσιάσει αντίφαση στον εαυτό του. Τι να πω, σας βγάζω το καπέλο, πώς το καταφέρνετε. Ε, Επίση, πολλοί μπήκαν, διάβασαν τη δήλωση και έφυγαν. Υποθέτω ότι κάθονται στα γραφεία τους και ελπίζω να διαβάζουν το κείμενο για το οποίο εκλήθησαν να μιλήσουν, γιατί ίσως δεν το είχαν διαβάσει προσεκτικά. Ε, να δούμε το θέμα της προστασίας των διπλωμάτων. Αυτό το πακέτο δεν μιλάει για απονομή των διπλωμάτων. Αυτό δεν υπάρχει στο 118, πρόκειται για την προστασία των διπλωμάτων. Κάποιο διπλωμά δεν απενεμήθηκε, διατηρείται και ένα το οποίο απενεμήθη μπορεί να μην μπορεί να διατηρηθεί. Ε, για να μπορέσει κανείς να επικαλεστεί προστασία πρέπει να προσφύγει σε 25 κράτη. Τώρα κάνει μία προσφυγή. Όποιος λέει εδώ ότι ε, δεν ε, μειώθηκε το κόστος για τις μικρομεσαίες, ε, πραγματικά αυτό δεν είναι εύλογο. Ε, βεβαίως και βοηθούνται οι μικρομεσαίες. Επίσης, όταν λέμε ε, για τις συζητήσεις μεταξύ επιστημόνων στην επιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα. Ε, πραγματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν ε, σε τέτοια θέματα δεν αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εμείς διασώσαμε τη θέση του δικαστηρίου στις προδικαστικές ε, ε, αποφάσεις. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο. Αυτή εξ αρχής δεν ήταν άλλο το αντικείμενο. Και σας λέω, ποιο είναι σήμερα κατά του πακέτου και ψηφίσει κατά του πακέτου, παίζει το παιχνίδι των μεγάλων παίζει το παιχνίδι των μεγάλων επιχειρήσεων ενάντια στις μικρομεσαίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ε, Ραπκάη. Ευχαριστώ όλους κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι τρεις εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνία θα τεθούν σε ψηφοφορία σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Και η συνεδρίασή μας διακόπτεται μέχρι τις 12. Σας ευχαριστώ πολύ.